Can we start, please? We are already late and uh, not having too much of... Να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε ήδη αργήσει. Ε, λίγα μέλη είναι παρόντα, αλλά μπορεί να μείνουν και λιγότερα αν δεν αρχίσουμε. Οπότε εγώ αντικαθιστώ εδώ κάποιον ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τάξης 3. Σας καλωσορίζω όλους εδώ σε αυτή την ακρόαση Τη ακροαση Tax 3. Σήμερα θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα μέρο του οικονομικού έργου που μα έχει ζητηθεί. Ε, οι μελέτε αυτέ είναι μια ένα σημαντικό μέρο ε, της δουλειάς ε, παίρνουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Έχουμε τρία ζητήματα που θα εξετάσουμε σήμερα. Πρώτα, ε, τα χρυσά διαβατήρια και τα χρυσέ θεωρήσει, ε, το, ο κίνδυνος Ε, ε, στη ε, στο και στις λιμένες και ακόμα ένα θέμα να σας πω ότι την Δευτέρα είχαμε μια ακρόαση για τις χρυσές βίζες, τις χρυσές θεωρήσεις και ε, ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι που είναι εδώ μαζί μας για το πρώτο ζήτημα η κυρία Αμαντίν Ζερά η οποία θα μας παρουσιάσει την δική της μελέτη, τη μελέτη του συναδέλφου της της συναδέλφου της Τσελοντή Τυριών για το θέμα ακριβώ των Golden Visas και των χρυσών διαβατηρίων. Ε, μας έλειπαν και κάποια στοιχεία αριθμητικά τη Δευτέρα. Ε, λοιπόν, ε, παρακαλώ μπορείτε να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλό απόγευμα σε όλους. Όπως θα γνωρίζετε, οι χρυσέ θεωρίες και τα χρυσά διαβατήρια είναι ένα έτσι, πολύ καυτό θέμα, ένα θέμα επικαιρότητα. Σε αυτή τη ε, διαφάνεια μπορείτε να δείτε πώς αυτό το ζήτημα ε, εμφανίζεται στα προσέλιδα των εφημερίδων. Ε, μόνο σε χθεσινά είναι αυτά που βλέπετε. Η Ελλοντή και εγώ λοιπόν χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση όλες οι ιστορίες που έχουμε ακούσει για την ηθαγένεια και την άδεια παρα, παραμονής έχουν ε, ρίξει το φως στην περίπτωση αυτή. Μιλάμε για διαφθορά, ξέβλημα χρήματος, σύγκρουση συμφερόντων. Από ό,τι φαίνεται όσο περισσότερο μαθαίνουμε ε, για αυτά τα προγράμματα ε, όλο και πιο σκοτεινά είναι. Δημιουργείται μεγάλη σύγχυση και δεν ξέρουμε τελικά ακριβώ για ποιο πράγμα μιλάμε. Α διευκρινίσουμε καταρχήν λοιπόν κάποια πράγματα. Στη μελέτη μας εμείς επικεντρωθήκαμε σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με επενδυτέ ε, που δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που έρχονται με μία τιμή. Ε, δεν μιλάμε δηλαδή για προγράμματα που δεν έχουν ελάχιστα ποσά, που δεν είναι οι κλασικές θεωρήσεις ε, τύπου επιχειρηματιών. Επίσης ε, δεν αναφερόμαστε ε, στην ηλεκτρονική διαμονή, στην εικονική διαμονή που υπάρχει σε ένα κράτος μέλος. Επίσης δεν μιλάμε ε, για την απόκτηση ηθαγένειας με βάση κάποια συγκεκριμένα επιτεύγματα. Αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα βέβαια σε επίπεδο διαφάνειας, αλλά εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι κλασικές περιπτώσεις ε, χορήγηση ηθαγένεια λόγω κάποια επένδυση. Για να μην υπάρχει λοιπόν καμιά σύγχυση, να το πούμε πολύ απλά, αυτά που καλύπτει η έρευνά μα είναι τα εξή. Σε ανταλλαγή, σε αντάλλαγμα μια σημαντική επένδυση, δίνονται δικαιώματα ηθαγένειας ή παραμονής. Και αυτό το προβλέπει η νομοθεσία. Είναι πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο και στα μίντια για αυτά τα προγράμματα και ορισμένε φορές δημιουργείται σύγχυση και ορισμένε φορές μάλιστα είναι αντιφατικέ πληροφορίες. Για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακριβή τα στοιχεία μα, βασιστήκαμε μόνο σε επίσημα έγγραφα. Πριν όμω περάσουμε στι λεπτομέρειε των προγραμμάτων αυτών, θέλουμε να διευκρινίσουμε ένα ακόμα στοιχείο, μια και συχνά ακούμε ότι αυτά τα προγράμματα ε, είναι ουσιαστικά ένα μια πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το να λάβει ε, κάποιο ε, μια άδεια παραμονή σε ένα κράτο μέλο δεν δίνει δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια με τη ηθαγένεια. Υπάρχει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Έχουν πολύ διαφορετικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, το να λάβει κάποιο μια διαπαραμονή σε ένα κράτο μέλο τη Ένωση δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει το δικαίωμα να ε, μείνει να διαμείνει οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να έχει κάποιο δικαίωμα να, να ζήσει οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει ο υπήκο τρίτη χώρα να έχει φύγει από το κράτο μέλο τη Ένωση για περίοδο 5 ετών. Και κάποια προγράμματα δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του ατόμου, οπότε δεν πληρείται συγκεκριμένη προπόθεση. Από τη στιγμή που διευκρινίσαμε λοιπόν αυτό, ε, διαπιστώσαμε ότι 18 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν τέτοια προγράμματα ε, άδειε παραμονή με βάση συγκεκριμένη επένδυση. Τέσσερα κράτη-μέλη εξ αυτών ε, έχουν επιπλέον ε, και προγράμματα χορήγηση ηθαγένεια πέρα από την άδεια παραμονή. Εξετάζοντα τι λεπτομέρειε όλων των πραγμάτων αυτών όμω, είδαμε ότι υπάρχουν πολλέ παραλλαγέ. Πρώτον, η φύση και το ποσό τη επένδυση απικύλει σε μεγάλο βαθμό από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε προσωρινέ άδειε παραμονή, αλλού μόνιμε άδειε παραμονή, αλλού ηθαγένεια. Κάποια ζητούν φυσική παρουσία στο έδαφος, αλλά όχι. Και τώρα θα πάμε λίγο πιο βαθιά στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Ε, για να γίνουν κατανοητές όλες ε, οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων, εξετάσαμε αφενός την υποχρέωση, τις υποχρεώσεις που έχει ο ετών και αφετέρου τα δικαιώματα που τη χορηγούνται ε, ως αντάλλαγμα. εξηγούνται βεβαίως όλα τα, όλες οι μεθοδολογικές επιλογές μας ε, και όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε. Αλλά να σας πω εν συντομία ποια είναι τα βασικά κριτήρια που αποκολουθήσαμε στη μελέτη μας. Εγκρίναμε μια σειρά από κριτήρια που σχετίζονται πρώτα με τις ε, προϋποθέσεις πρόσβασης. Εξετάσαμε εδώ τις υποχρεώσεις επένδυσης και, τη, και την απέτηση φυσικής παρουσίας. Το δεύτερο σετ δεδομένων εξετάζει το κριτήριο της ε, των πλεονεκτημάτων αυτού του καθεστώτος, πρόσβαση στην κινητικότητα, καθώς και κάποια ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Όπως βλέπετε, εδώ λάβαμε υπόψη μας ε, ένα, ένα, ένα ζήτημα που ανησυχεί ιδιαίτερα τη δική Επιτροπή, τη φορολογική διάσταση, κάτι που δεν καλύπτεται συχνά σε άλλες εκθέσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό, σε άλλες μελέτες. Εδώ βλέπουμε σε αυτό τον πίνακα, ε, ο, συνδυάσαμε όλα τα κριτήρια. Όπως μπορείτε να δείτε, ελπίζω, αυτή η μεθοδολογία μας έχει επιτρέψει να δούμε ποια είναι τα προγράμματα που έχουν τις μικρότερες απαιτήσει ε, με τα υψηλότερα δικαιώματα. Τα βλέπετε εδώ πάνω δεξιά. Στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στη Λετωνία, στη Μάλτα και στην Πορτογαλία συμβαίνει αυτό. Θέλω, να είμαι σαφής εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα προγράμματα δημιουργούν ζητήματα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διαφάνειας. Όμως, ο στόχος μας ήταν να συνδυάσουμε πολλά και διάφορα κριτηρία μεταξύ των οποίων αυτά που αφορούν και, τη φορολόγηση, και στη φορολόγηση. Ε, τα προγράμματα αυτά έχουν τα εξή κοινά. δεν απαιτούν φυσική παρουσία ή πολύ, πολύ μικρή. Οι περισσοτερε επενδύσεις είναι παθητικής υφής και είναι συνήθως χαμηλά συνήθως μπορεί να είναι απλά η αγορά, το ποσό μιας Porsche ή μιας Ferrari ε, μεταχειρισμένης. Δίνονται λοιπόν άδειε παραμονής ε, ε, στις χώρες αυτές και αλλού δίνονται, δίνονται και ηθαγένεια προς στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στη Μάλτα. Επίσης η πρόσβαση σε, η πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα σημαίνει και πρόσβαση σε φορολογικό ευνοϊκό σύστημα. λιγότερο από 20% φορολόγηση ε, προσωπικού εισοδήματος στην Εσθονία και στη Λετωνία. Επίσης στην Κύπρο, Ιρλανδία, Μάλτα και Πορτογαλία ε, υπάρχει ε, ένα καρποκόμι ποσό 100.000 ευρώ για τα ξένα εισοδήματα. Στην Ιταλία εξαιρώνεται εντελώ τα ξένα εισοδήματα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι στη Λετωνία 40% όλων των άδειων παραμονής χορηγήθηκαν μέσω αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή επένδυση για ε, ε, ε, ε άδεια παραμονής. 50% όλων των χορηγήσεων ηθαγένεια στη Μάλτα επίσης προέρχονται από αυτά τα προγράμματα. Στη μελέτη μα βεβαίω αναλύσαμε λεπτομερώ μια σειρά από στοιχεία που αφορούν τα προγράμματα αυτά. Εμεί θέλουμε να επικεντρωθούμε όμω σε δύο στοιχεία εδώ. Πρώτον, το θέμα του κινδύνου που συνοδεύει αυτά τα προγράμματα και το δεύτερο είναι ο οικονομικός αντίκτυπος. Πρώτα απ' όλα ο κίνδυνος. Όπως όλοι γνωρίζετε, η έλεγχη για την ακαιρεότητα των προγραμμάτων ε, για τους ετώντες και που προέρχονται τα χρήματα είναι κάτι το οποίο ε, αμφισβητείται σημαντικά. Πρέπει εδώ να πούμε ότι ζητήματα που σχετίζονται υποθέσει μάλλον που σχετίζονται με αυτά τα προγράμματα έχουν οδηγήσει ε, σε έρευνε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί ότι αυτά τα προγράμματα είναι εξαιρετικά ευάλωτα ε, και σε διαφθορά. Όλα αυτά τα ζητήματα πλέον στοιχειοθετώνται. Κάτι που θα θέλαμε να αναφέρουμε κάπως πιο λεπτομέρως εδώ είναι ο κίνδυνος ό,τι αφορά την φορολογική διαφάνεια με αυτά τα προγράμματα. Αυτό είναι που σα απασχολεί και εσά όλο ιδιαίτερο. Είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των ατόμων που υποβάλλουν τέτοια αίτηση για φορολογικού λόγους, θα μπορεί, μπορεί όμως κανείς να πει ότι τα, κίνη, τα φορολογικά κίνητρα είναι ένα σημαντικός παράγοντας για τη ζήτηση τέτοιου είδου ε, προγραμμάτων. Πρόσφατα ο ΣΑΚ ξεκίνησε μια διαβούλευση για το βαθμό στον οποίο αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ε, για να παρακαμφθούν, παρακαμφθεί το CRS, ε, ε, τα κοινά πρότυπα αναφοράς δηλαδή. Ε, τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα από πλευράς φορολογικής ε, διαφάνειας και βεβαίως είναι και βάλωτα και σε ό,τι αφορά την, το δεχόμενο φοροδιαφυγής. Ε, επειδή δεν υπάρχει η υποχρέωση φυσικής παρουσίας, ο φορολογούμενος με το που λαμβάνει το δικαίωμα ηθαγένειας ή διαμονής μπορεί απλά ε, να, να φέρει κάποια κείμενα, να παρουσιάσει κάποια κείμενα ε, διαμονής για να έχει και φορολογική έδρα στη χώρα αυτή χωρίς να έχει βάλει το πατήσει το πόδι του εκεί. Πέντε από τα προγράμματα αυτά επίσης δίνουν στον επενδύτη τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ένα συγκεκριμένο ειδικό φορολογικό καθεστώ όπου έχει ε, φοροαπαλλαγή για το ξένο εισόδημα. Εδώ βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα για τις φορολογικές αρχές. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αυτό στην Κύπρο, μια χώρα που συμμετέχει στο CRS αλλά που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες ε, σε μια βάση αμοιβαιότητας. Εδώ θα θέλαμε να επιμείνουμε στο γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανταλλαγή πληροφοριών, διότι δεν είναι σημαντικό αυτό μόνο για να αποφύγουμε τη διπλή φορολόγηση, είναι σημαντικό και για να αποφύγουμε τη μη φορολόγηση. Να περάσουμε τώρα στον αντίκτυπο αυτών των προγραμμάτων θα αναφερθούμε στον οικονομικό αντίκτυπο σε επίπεδο κρατών μελών κυρίω. Βεβαίω στη μελέτη καλύπτουμε και τον κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο. Ε, δεν μπορεί κανεί να αρνηθεί ότι αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί σημαντική ε, συνεισφορά ε, βραχυπρόθεσμα στα δημόσια οικονομικά. Σε κάποια κράτη-μέλη αυτά τα προγράμματα δημιουργήθηκαν ακριβώ για να μπορέσει να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση. Όμω, πιο μακροπρόθεσμα, τα ωφέλη από αυτή την επένδυση είναι αρκετά αβέβαια. Πρώτα απ' όλα, όπως υπόθηκε νωρίτερα, δεν υπάρχει υποχρέωση για τον νέο ε, διαμένοντα ε, να διαμένει πραγματικά στη χώρα ή να, είναι φορο, ή να φορολογείται εκεί. Έτσι λοιπόν ο βαθμός στον οποίο αυτή η να ειναι να φορολογειται εκει ετσι λοιπον ο βαθμος στον οποιο αυτη η επενδυση ε, αυξάνει τη φορολογητέα βάση είναι σχετικός. Επίσης τα προγράμματα που καλύψαμε δεν απαιτούν απαραίτητα, δεν οδηγούν απαραίτητα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για θέλουν να δώσουν μια όθηση ε, στον τομέα παραδείγματο χάρη των κατασκευών, σίγουρα αυτό δημιουργεί και θέσει εργασία, αλλά δημιουργείται και πίεση στην αγορά κατασκευών και μπορεί να δημιουργηθεί επίση και μια φούσκα κερδοσκοπική στο συγκεκριμένο κλάδο. Επίση, αν ένα κράτο μέλο ε, βασίζεται υπερβολικά στι οικονομικέ ροέ που θα προκύψουν τα προγράμματα αυτά, από εκεί πέρα είναι βάλωτο εφόσον ε, σταματήσει αυτή η ροή. Και μακροοικονομικά δεν θα είναι και τόσο ανθεκτικό Δηλαδή μπορεί αυτό, αυτό το χρυσορυχείο να γίνει ναρκοπαίδιο. Ε, και έχουμε δει πολύ διφορούμενα αποτελέσματα στο αφορά τα ωφέλη αυτών των προγραμμάτων μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα τελειώνοντα να αναφερθώ στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ πρώτη όψεω θα μπορούσε κάποιο να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα εδώ. Όμω η νομική αρχή της, ε, ε ε, ειλικρινούς συνεργασίας ε, δημιουργεί ένα θέμα, ιδιαίτερα για τη χορήγηση ηθαγένειας. Ε, υπάρχουν κάποια ρίσκα εδώ. Έτσι λοιπόν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χορήγηση ηθαγένειας σαν κράτος μέλος ε, δεν είναι χωρίς επιπτώσει για το σύνολο τη Ένωση σύνολο και υπάρχουν διάφοροι τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Πρώτον, το πλαίσιο για την καταπολέμηση του εξελίγματο χρήματο είναι ήδη αρκετά ισχυρό ε, έχει αναγνωριστεί ο κίνδυνος αυτών των προγραμμάτων στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Οδηγίας που και η μεταφορά της οδηγίας αυτής έως τον Ιανουάριο 2020 θα είναι ένα σημείο κλειδί. Η Κομισιόν θα μπορούσε λοιπόν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των κρατών μελών και της επαγρύπνησής τους ε, σε ό,τι αφορά τους ετούντες. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει όπως και στα πλαίσια της έρευνας που έλαβε χώρα στη Μάλτα από τις Ευρωπαϊκές Τραπεζικές Αρχές. Δεύτερον, πάντα στα πλαίσια της φορολογικής διαφάνειας θα μπορούσε η Κομισιόν να ζητήσει να προτείνει βέλτιστες πρακτικές με βάση τους κανόνες του ΟΣΑ και τα κοινά πρότυπα αναφοράς. Στις γραμμές του ΟΣΑ ε, λέγεται ότι η κατάχρηση του CRS μπορεί να αποφευχθεί εφόσον εφαρμοστούν σωστά οι διαδικασίες επαγρύπνησης, να υπάρχει ε, μια προσέγγιση που θα βασίζεται στο συστημικό κίνδυνο. Είναι και αυτό ε, μια πρόταση. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει προστασία των whistleblowers σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι συχνά παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο για να μπορέσουν να αποκαλύψουν τέτοιες υποθέσεις. Επίσης χρειάζεται ένα πλαίσιο ε, μιας διακυβέρνησης που να λογοδοτεί για να είναι βιώσιμη και να είναι και αξιόπιστη, να έχουν και καλή φήμη αυτή η, αυτά τα προγράμματα. Χρειάζεται συλλογή δεδομένων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο για την αξιοπιστία και τη διαφάνεια, αλλά και για να μπορούμε να αξιολογήσουμε από εκεί και πέρα ε, τα προγράμματα αυτά. Όπω και να έχουν τα πράγματα, και αυτό είναι το τελευταίο μα σχόλιο. Εάν παραμείνουν αυτά τα προγράμματα χορήγηση ηθαγένεια και άδεια παραμονή, τα, οι στόχοι των οικονομικών ωφελών πρέπει να ιδωθούν ε, σε απόλυτη συνάρτηση με τους κινδύνους ε, που, που ελοχεύουν. Συχνά μπορεί να θεωρηθεί παρέκκληση από τους ε, παραδοσιακούς παραδοσιακούς οδούς μετανάστευσης, οπότε εδώ δημιουργούνται διακρίσεις. Πρέπει να παραμείνει λοιπόν η εμπιστοσύνη και το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαστε διάθεσοι για να απαντήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Και πριν ε, προχωρήσουμε, να ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Τάξε, ως εισηγητή από πλευράς του ΕΛΚ, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να κάνω και κάποια σχόλια. Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ποια είναι τα ωφέλη του προγράμματος αυτού για τις χώρες. Το μοναδικό, οι μοναδικοί που ωφελούνται είναι οι εταιρείε κατασκευαστικέ. Σε ό,τι αφορά δηλαδή και τις τιμές που πουλάνε στη συνέχεια τα έργα τους στους αλλοδαπούς. Αλλά να σας πω ότι τέτοια προγράμματα εξακολουθούν να υφίστανται γιατί δεν μπορούν να υπαρχούν σε οποιαδήποτε σωστή οικονομική αξιολόγηση. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να δώσω την αντιπροεδρία, την προεδρία μάλλον στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Τάξα. Thank you very much. And I must um, start by... Σας ευχαριστώ. Να σας ζητήσω συγγνώμη και όλος ιδιαίτερος από τους προσκεκλημένους μας, αλλά και από τη γραμματεία δικό μου το σφάλμα. Είχα χρόνο και σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι που με αντικαταστήσατε. Για να μην καθυστερήσουμε λοιπόν τώρα, να δώσουμε το λόγο στην επόμενη ομιλητρία. Ε, I'm sorry, with the transition Ναι, συγγνώμη. Έχουμε καταρχάς να δώσουμε το λόγο για να απαντήσει η ομιλητρία στην ερώτηση του κ. Νίτερμαγερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στην μελέτη, όντω προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε τον οικονομικό αντικτύπο και ενδεχόμενο όφελος από πλευρά των επενδύσεων των κρατών μελών σε πόσο σωστό ΑΕΠ. Άρα μιλάμε για 9,2 δισεκατομμύρια εισρωές της ε, οικονομίας των κρατών μελών. Δεν μπορέσαμε ωστόσο να αξιολογήσουμε κατά πόσο αυτές οι επενδύσεις θα γίνονταν έτσι κι αλλιώς και χωρίς τα προγράμματα αυτά δηλαδή. Έχουμε λοιπόν κάποια αριθμητικά στοιχεία, δεν μπορούμε όμως να αποφανθούμε κατά πόσον αυτές οι επενδύσεις έγιναν μόνο λόγω της ύπαρξης ακριβώς του προγράμματος. So, Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Φαντεκάντελάρα τώρα έχει το λόγο. Δεν είναι παρόν. η κυρία Νίνα Γκίλ. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίασή σας. Είναι ευρέως δεδομένο το φαινόμενο αυτό, το οποίο το παρουσιάσετε πολύ α, επιτυχημένα. Ο συνάδελφος λίγο έφρυξε με τα στοιχεία που μας δώσατε και οι μαρτυρίες ε, που έχουμε λάβει είναι παρόμοιες, ότι παντού στην Ευρώπη έχουμε 6.000 νέους πολίτες και περίπου 2.000 νέους κατοίκους που προέρχονται από το σύστημα, αυτό το πρόγραμμα για τις χρυσές θεωρήσεις ε, τα τελευταία χρόνια αυτό. Και τα κράτη-μέλη προσελκύουμε τον τρόπο αυτό 25 δισεκατομμύρια δαπέ επενδύσει. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν μπει σε ένα εσωτερικό ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά την παροχή αυτή ηθαγένεια, άδεια παραμονή κτλ. Ενώ εκ παραλίλου, κοιτώντα ε, το πρώτο θέμα που μας απασχολεί, που απασχολεί το κοινό, είναι οι πρόσφυγες. Φαίνεται ότι έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά. Για άμα είναι κανείς μετανάστης, ε, πρέπει να περάσει τεστ, ε, δοκιμές, ε, ενώ άμα έχει λεφτά, μπορεί κανείς να αποκτήσει ηθαγένεια χωρίς κανένα από αυτά τα προβλήματα. Γιατί υπάρχει αυτό το διπλό σύστημα. Για την Επιτροπή λοιπόν υπάρχουν ανησυχίες. Δεν είμαι κατά του να προσελκύουν τα κρατημέλη αλλά τα πες επενδύσεις. Μην με παρεξηγήσετε. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά και ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών. Κάποια κρατημέλη εξαρτώνται, εξαρτώνται μάλιστα πολύ σοβαρά από τα προγράμματα αυτά. Θα μπορούσε αυτό να προκαλέσει οικονομική αστάθεια. Δεν το γνωρίζω και θα ήθελα να μου πείτε από πλευρά τη έρευνά σα τι προέκυψε. Τέτοια ζητήματα οικονομική αστάθεια. Και επίση. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στις τιμές των ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη χώρα μου. Πολλά από αυτά τα άτομα που έχουν έρθει με βελτιωμένες τέτοιες θεωρήσεις αγοράζουν προφανώς ακίνητα σε πολύ ψηλές τιμές, αλλά αυτό προφανώς και επηρεάζει και τις τοπικές τιμές. Και τελικά ο κόσμος, ο κόσμος της χώρας δεν μπορεί να πληρώσει το ακίνητο που θα ήθελα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη συνέχεια σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που επικράτει προ το νομικό σύστημα και το καθεξή. Η έρευνά σα εξέτασε και αυτού του τομεί. Κάντε κάποιε συστάσει ε, για το πώ θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσω της δέουσας επιμέλεια, αλλά πείτε μου αν ε, στην έρευνά σα πραγματεύεστε και αυτό το στοιχείο. Να απαντήσω την ερώτησή σας και η Ελλοντή θα απαντήσει όσα δεν θα σας απαντήσω εγώ. Σε ό,τι αφορά τον παραλληλισμό με την ε, προσφυγική κρίση, προφανώς και το θέσαμε αυτό στην μελέτη. Υπάρχει το αίσθημα διακριτικής ε, μεταχείρισης. Ε, γιατί συνήθως οι διαδικασίες αυτές είναι πιο εύκολες, πιο γρήγορες. Η οικογενειακή επανένωση είναι πολύ πιο εύκολη μέσω του προγράμματος σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα που επικρατούν για τις πρόσφυγες. Άρα μας απασχολεί αυτή η αίσθηση διακριτικής μεταχείρισης που προκαλεί προφανώς και δυσαρέσκεια και έλλειψη εμπιστοσύνη από τον πολίτη. Μία έρευνα έγινε στη Μάλτα και μία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι δύο καταδεικνύουν ότι οι πολίτες είναι κατά των προγραμμάτων επί της αρχής. Δεν εγκρίνουν ούτε τη φύση ούτε την ε, φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών. Άρα υπάρχει και κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπο. Το αναφέρουμε αυτό στην ε, έρευνα. Για τον οικονομικό τώρα αντικτύπο να δώσω το λόγο στην ελλοντή για να το σχολιάσω. Ναι, όντω, στην ε, έρευνα εξετάσαμε το μακροοικονομικό αντικτύπο και εδώ βασιστήκαμε σε μία μελέτη IMF η οποία όντως τονίζει ότι υπάρχουν αντίκτυπος από αλλαγή του, της πολιτικής σε ό,τι αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική αστάθεια και διακυμάνσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αντίκτυπο για τις τιμές των ακινήτων, εδώ δυσκολευτήκαμε να βρούμε τα αριθμητικά στοιχεία, γιατί είναι αματοποιημένα σε επίπεδο κρατών μελών και δεν υπάρχει συγκεκριμένη... συγκεκριμένος καταμερισμός. Όντω, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία και στην Κύπρο προέκυψε ότι υπήρξε αύξηση στις τιμές των ακινήτων και στη Μάλτα, με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένω. Και αυτό προφανώς επηρεάζει τους πολίτες της Πορτογαλίας και της Κύπρου σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά κινητών. Η Πρόεδρος. Ο κύριος Νίλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία μικρή ιστορική αναδρομή να κάνω. Στη Φιλανδία υπήρξε εισρωή Ρώσων πολιτών τη δεκαετία του 90 γιατί αισθάνθηκαν, αισθάνονταν δικαίω κάπως ανασφαλείς στη χώρα τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ε, γνωστός μουσικός ε, τσελίστας, ο κ. Μαστραφοπόβιτς. Αυτό που έγινε λοιπόν στη Φιλανδία πριν από μία μήνα ήταν διαφορετικό. Μία αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας έλαβε χώρα σε τμήμα της Φιλανδίας. Ένα τμήμα της Φιλανδίας που γενικά θεωρείται πολύ φιλήσυχο και φιλερινικό, το φιλανδικό αρχιπέλαγο. Και τελικά υπήρχε ένας τύπος ο οποίος είχε μια εταιρεία που φαινόταν γραμματοκιβωτίου και είναι πολλά τα νησάκια στην ε, στο δρομολόγιο του φέρει από τη Φιλανδία προς τη Σουηδία και ενδεχομένως αυτό να διαδραματίσει ρόλο κλειδί σε μια ενδεχόμενη κρίση. Όταν προέκυψαν λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία, αυτός ο τύπος είχε διαβατήριο Μάλτας. Και πριν από κάποιες εβδομάδες, πριν από κάποιους μήνες μάλλον, έγινε μια ακρόαση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για μαλτέζικες τέτοιες ε, ψευδοπιχειρήσεις. Και τότε λοιπόν έθεσα το ερώτημα των μαλτέζικων διαβατηρίων, ε, ερώτησα τότε στην ακρόαση, ήταν θέμα ευρωπαϊκό ή μαλτέζικο. Και τότε οι μαλτέζικες αρχές και οι εκπρόσωποι αυτών αρνήθηκαν να απαντήσουν, γιατί φυσικά είτε ναι έλεγαν είτε όχι, χαμένοι θα ήταν και έτσι δεν σχολίασαν ως συνήθως. Τώρα λοιπόν κατανοούμε το εξής. Αποδεχόμενα, αποδεχόμενα νέους πολίτες η αποδοχή μάλλον νέων πολιτών στην ε, Φιλανδία είναι θέμα τελειωμένο, είναι θέμα κρατών μελών. Έχει γίνει. Αν όμως υπάρχει η μου υποψία ότι υπάρχει κάποιο οποίο συνήθως είναι υπόβαθρο ή κάποια πρεστορία στη Ρωσία, το οποίο συνήθως είναι το ίδιο, ε, ε, ε, χρειαζόμαστε κανόνες. Η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών φαίνεται ότι δεν εξαγάγεται στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο. Ο καθένας κοιτάει τι πιστώσεις έχει και τι έχει δανειστεί, ο καθένας τα δικά του κοιτάνε τα λογιστικά αν θέλετε, δεν κοιτάνε όμως τη συνολική εικόνα. Και αν δεν ε, τα κοιτάξουμε όλα αυτά συνολικά, δεν θα μπορέσουμε να τα καταπολεμήσουμε. Τα αριθμητικά στοιχεία που μας αναφέρετε το ίδιο ακριβώς δεικνύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πανοραμική θεώρηση του προβλήματος. Ιδάλλως δεν θα καταπολεμήσουμε ποτέ την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πηγές, δεν θα καταπολεμήσουμε ποτέ την χρηματοδότηση της δημοκρατίας και άλλες τέτοιες μορφές εγκλήματος. Και πραγματικά θεωρώ ότι έχουμε κάποια πολύ πραγματικά προβλήματα ενώπιον μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σχολιάσετε, να απαντήσετε. Well, we, we have seen, I mean... Κοιτάξτε, το διαβάζουμε και στα νέα ε, κάθε μέρα ότι υπάρχουν διαρκώς τέτοιου είδους ε, κατηγορίες και υποψίες. Ε, φαίνεται όμως ότι τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει αρχίσει και ε, μελετά το θέμα ε, πολύ ζεστά και μάλιστα στη Μάλτα έχει ξεκινήσει έρευνα και τον Ιούλιο επεδείχθη ότι η Μάλτα έχει παραβιάσει τις απαιτήσει της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και αυτό απεδείχθη μετά από έρευνα Άρα καταλαβαίνουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλωστε το αποδεικνύει και η εργασία της δικής σας Επιτροπής ε, όπως και ε, στην Επιτροπή ΠΑΝΑ τα θέματα αυτά λαμβάνονται πλέον πολύ σοβαρά υπόψη ε, και βεβαίως έχουν και διασυνοριακό αναμφισβήτητο και αναμφίβολο στοιχείο και οπωσδήποτε έχουν και αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο κύριος Τάνκ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας ε, είπαμε πολλά ε, όσον αφορά την ανηθικότητα ας πούμε, αυτού του, εργαλείου, αυτού, του προγράμματος που, δεν, που είναι αντιδεοντολογικό. Ή, μάλιστα, πολλοί κόσμος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι άδικο αυτό το σύστημα και σίγουρα ε, μπορεί να υπάρξουν ε, όχι μονάχα ε, επιπτώσεις που αφορούν το ίδιο το κράτος που δίνει τη θεώρηση αλλά και, άλλες, και σε άλλες χώρες όσον αφορά φοροαποφυγή και ξέπλυμα χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων, παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε δε την αίσθηση ότι αυξάνεται αυτή η διαδικασία και δημιουργείται με τον τρόπο αυτό όλο και περισσότερο αυξανόμενη, ε, όλο και αυξανόμενος φορολογικός ανταγωνισμός. Εν πάση περιπτώσει όμως. Δεν κατάλαβα καλά. Ε, έχετε ε, βρει αποδεικτικά στοιχεία ότι η διαφθορά και το ξέπλυμα προωθούνται κατά κάποιο τρόπο από αυτό το πρόγραμμα. Έχετε συγκεκριμένα από το Clock Witness, από την ε, υπάρχει μαύρη λίστα του ΩΣΑ, ε, υπάρχουν πολλές υποψίες, αλλά εσείς βρήκατε κάποια συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, γιατί διαβάζω ε, ότι ε, στις, ε, στα, στα συμπεράσματά σας ότι η εφαρμογή της οδηγίας για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων ενδεχομένως παραβιάζεται. Επίσης, για μερικές χώρες το μέγεθος είναι σημαντικό γιατί διαφορετικά δεν θα συζητούσαμε για μικροοικονομικές εμπλοκές. Δεν ξέρω βέβαια πόσα μπορείτε να μας πείτε από όλα αυτά που έχετε βρει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τεριάν. Όσον αφορά το πρώτο που θίξατε, αναθεωρούμε, στην, μάλλον κάνουμε μια επισκόπηση όλων των ε, περιπτώσεων που επισήμως έχουν ε, ε διαρευνηθεί. Στη δικιά μας δεν αναφερόμαστε ε, σε πιθανές κατηγορίες υποψίες, αλλά σε συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει. Ε, όσον αφορά την σωστή υλοποίηση της ε, MD, AMLD, της νομοθεσίας για την νομοποίηση παρανόμενων εσόδων σε ενωσιακό επίπεδο, είναι γεγονός ότι εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στις σωστές διαδικασίες και την συνοχή με αυτές τις διαδικασίες ελέγχουμε έχουμε και τόσα συνέβησαν στην Εστονία ας πούμε, κατέδειξαν ότι ε, δεν εφαρμόζεται σωστά η διαδικασία ε, της ε, της δέουσας επιμέλειας. Και μάλιστα στο παράρτημα 3 της πέμπτης οδηγίας αναφέρεται ε, ρητά ε, στους κινδύνους που ε, προκύπτουν και απορρέουν από τα προγράμματα παροχής διαμονής και ηθαγένειας. Και βεβαίως εσείς όπως και η Κομισιόν πρέπει να μελετήσετε και να βρείτε τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο η ο μακροοικονομικός αντίκτυπος ε, πραγματικά είναι πολύ ισχυρότερος ε, σε μικρότερες χώρες, στη Λετωνία ας πούμε, το 1% του ΑΕΠ αντιπροσωπεύεται από αυτήν την διαδικασία, στην Κύπρο 2,5, δηλαδή πολύ παραπάνω από τη Γεωργία που είναι στο 1,3. Ε, αναφέρομαι σε συμβολή στο ΑΕΠ. Ναι, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποχρέωση ε, ε, διαμονής στην χώρα, πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε ποια είναι η, ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος στη φορολογική κατάσταση. Είπατε όμως ότι δεν έχετε δηλαδή τον αντίκτυπο στον κυβερνητικό Προπολογισμό. Ε, όχι, έχουμε είναι η απάντηση τα στοιχεία όσον αφορά τι επενδύσει, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το spillover ε, στην ε, συνολική οικονομική κατάσταση. Εδώ και εννέα χρόνια Εδώ και νέα χρόνια είμαι μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τέτοια είδου υποδοχή ε, δεν είχα ξαναζήσει σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι μπορώ να σας μιλήσω, ότι μιλάω και λέω αγαπητοί προσκεκλημένοι, αλλά όχι αγαπητοί σύντροφοι, ε, γιατί δεν έχουμε εδώ συναδέλφους. Ε, τι κρίμα και ό,τι σημαίνει αυτό και για την δημοσιότητα. Ήμουν συντονιστή και στην τάξη 1 και τάξη 2 και τάξη 3 ότι μιλάμε για 18 από τα 28 κρατημέλη που έχουν τέτοιε ε, ρυθμίσει, τέτοια προγράμματα. Δεν το φανταζόμουν αυτό ποτέ. Νόμιζα ότι ήταν κάποια φυσικά τα κρατημέλη, αλλά 18 από τα 28 είναι σαφώς πλειοψηφία. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για ένα φαινόμενο κατεξαίρεση. Μιλάμε για κάτι που έχει κατοχυρωθεί. Το θέμα αυτό Τα υπόλοιπα, 10 χρο... τα υπόλοιπα αυτά 10 κράτη-μέλη που δεν έχουν τέτοια προγράμματα το θέτουν ως πρόβλημα. Το συζητάνε. Έχω διάφορα ε, στοιχεία και τεκμήρια. Υπάρχει κάποια συζήτηση και κάποια διαφωνία και κάποια αντιπαράθεση μεταξύ των χωρών που προσφέρουν τέτοια προγράμματα και μεταξύ αυτών που δεν προσφέρουν τέτοια προγράμματα. Και κατά δεύτερον, δεύτερη ερώτηση, έχετε κάποια αριθμητικά στοιχεία, έχετε κάποια εντύπωση, πόσα άτομα εντός των κρατών μελών ε, είναι ουσιαστικά πολίτες από άλλα κρατημέλη. Υπάρχει το τελικό παράδειγμα για την ε, αλλαγή του αποκατοικίας. Για πόσα άτομα μιλάμε που χρησιμοποιούν αυτές τις εσωτερικές ε, διαδικασίες και τι ποσοστό και εδώ είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ποιες χώρες πόσοι έρχονται από πόσες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Thank uh, Λοιπόν, ακούστε, πρώτα απ' όλα είναι 18 τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν προγράμματα χορήγησης πάθεια διαμονής με αντάλλαγμα επενδύσεις. Θέλει όμως προσοχή, διότι κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μάλλον, ε, δεν είναι απαραίτητα επιχειρηματίες, δηλαδή... Ε, δεν είναι πάντα ενεργέ επενδύσει επενδύσεις, καθημερινή διαχείριση μιας επιχείρησης. προσπαθούμε να, πραγματικά να λάβουμε υπόψη αυτή, αυτή την ιδιαιτερότητα. 18 λοιπόν κράτη-μέλη με, με αντάλλαγμα ένα συγκεκριμένο ποσό επένδυσης, αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για παθητικέ ε, επενδύσεις, δεν αφορούν παραδείγματος χάρη όλα τον τομέα τον κατασκευαστικό ή των ακινήτων, ε, εξαρτάται σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Στο παράτημα 1 και 2 πάντως εμείς εξηγούμε επακριβώς και στις λεπτομέρειες ε, τι έχουμε κάνει. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα συμπεριφορά και το τι συμβαίνει στο Συμβούλιο, για να είμαι ειλικρινή, εγώ δεν έχω, δεν έχω απάντηση στο ερώτημά σα. Και σε ό,τι αφορά τα μέλη, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα προγράμματα αφορούν μόνο μη Ευρωπαίους πολίτες, μόνο υπηκόους τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα, ναι, αλλά τα φορολογικά κίνητρα, τα φορολογικά πλεονεκτήματα δεν συνδέονται απαραίτητα με το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι προσβάσιμα και για Ευρωπαίους πολίτες που θα μπορούσαν να έχουν, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία, ε, τη φορολογική του έδρα. Ε, ή στην Πορτογαλία, η ίδια περίπτωση. Ε, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ε, να, έχει, να, διαμένει στην Πορτογαλία μέσω του προγράμματος αυτού για να έχει να συμμετέχει στο φορολογικό πρόγραμμα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις αιτήσει και τα ποσοστά επιτυχών αιτήσεων εκτός ενώσης, ε, για το CBI μιλάμε για πάνω από 5.000 πολίτες τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ηθαγένεια αυτό και την άδεια παρα... παραμονής 126.000 άνθρωποι τα τελευταία πέντε χρόνια είναι συντηρητικές αυτές οι εκτιμήσεις όμως γιατί βασίζουμε τα στοιχεία αυτά μόνο στα ε, διαθέσιμα στοιχεία από επίσημες κυβερνητικές πηγές ε, γι' αυτό και διαφέρουν σε σχέση με αυτά που θα ακούσετε αλλού. Αυτά πάντω είναι τα επίσημα στοιχεία, οπότε αναγκαστικά είναι ε, και πολύ συντηρητικά, μια και πάνω τα μισά κράτη-μέλη δεν δημοσιεύουν καθόλου τέτοια στοιχεία. Τώρα έχω και εγώ κάποιε ερωτήσει, λέει η Πρόεδρος, να πω ότι στη δική μου χώρα, στην Πορτογαλία, όπου υπάρχει αυτό το προτιμησιακό φορολογικό καθεστώ για του Ευρωπαίου πολίτε, αυτό είναι εκτό των χρυσών θεωρήσεων αλλά είναι και αυτό ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών της Τρόικα, έτσι. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές, Τρόικα. Ε, και βέβαια ε, δεν ε, επανεφεύραν τον τροχό, αντιγραφή είναι και αυτό. Κάποια κρατημέλια έχουν αρχίσει να ξυπνάνε, επιτέλους ίσως να ξυπνάνε οι πολίτες τους, αλλά εγώ έθεσα, έθεσα πολλά ερωτήματα στην Κομισιόν τόσα χρόνια. Πώς επιτρέπεται αυτό. Διότι πρόκειται για σαφή διάκριση σε βάρος των υπηκών της χώρας μου. Διότι αυτοί πλήρωναν τους φόρους τους. Πολύ υψηλότερου Ενώ δίναμε φοροαπαλλαγές σε Γάλλου, Βρετανούς, ε, Σουηδούς για να διαμένουν στην Πορτογαλία. Και αυτό γίνεται με σοσιαλιστική κυβέρνηση. Και λυπάμαι που το λέω και ρώτησα τον κύριο Σεντένο που είναι και πρόεδρος του Eurogroup αν πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Τώρα για τι χρυσές θεωρήσεις, το ερώτημά μου είναι το εξή. Ένας από τους λόγους στι συστάσεις σας ε, ε, αναφέρεστε στο θέμα ε, της παρακολούθησης. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει δημοσιο, δημοσίευση ε, των ετών, τουλάχιστον αυτών που, των δικαιούχων. Και αυτό σε μια χώρα όπως η Πορτογαλία ε, απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Γίνεται στη Μάλτα και στην Κύπρο. Αλλά στην Πορτογαλία δεν γίνεται. Και ε, <laughs> αυτό που είναι εξοργιστικό είναι ότι η αιτιολόγηση που δίνεται είναι τα, η, προσωπ, η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βεβαίω ε, άλλα κράτη-μέλη τα δημοσιεύουν. Και βεβαίω δεν είναι μόνο το θέμα των δικαιούχων. Είναι και για τα μέλη της οικογενειακής επανένωσης, για τους οποίους ισχύει παρεμφερές πρόγραμμα στην Πορτογαλία. Από το 2012 έχουν πάνω από 6.000 δικαιούχους ε, Golden Visa, αλλά πάνω από 11.000 μέλη οικογενειών του δικαιούχου έλαβαν άδεια παραμονής. Και αυτός είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος για να έρθουν διάφοροι έτσι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμφιβόλου ποιότητα. Αναφερθήκατε στην πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξυπνήματο χρήματο και εμεί εκεί, το Κοινοβούλιο δηλαδή, μπόρεσε να συμπεριλάβει μια αναφορά στην ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στην περίπτωση των χρυσών θεωρήσεων και των παρεμφερών ε, προγραμμάτων. Όμω, καθώ ε, αναφέρει και η έκθεση του Transparency International αυτό αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή την υποχρέωση δηλαδή ε, της, ε, αυτή η υποχρέωση της ε, δέουσας επιμέλειας. Το κάνουν οι τράπεζες σε έναν βαθμό, όμως οι δικηγόροι δεν το κάνουν. στον τομέα των ακινήτων δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όταν πήγα στην Πορτογαλία ε, στα πλαίσια του Panama Papers μας είπαν ότι δεν είχαν στοιχεία, δεν είχαν STR. Από αυτήν την πραγματική φάμπρικα που έχει δημιουργηθεί, έτσι. Ε, πώς βλέπετε εσείς ε, την ανάγκη αυτή ε, να πούμε ότι αν ένας ιδιωτικό φορέας υποχρεούται σε δέουσα επιμέλεια, πώς γίνεται η κυβέρνηση ε, ή ο κυβερνητικός φορέας που χορηγεί αυτή την άδεια παραμονής δεν υποχρεούται ε, να έχει αυτές τις ενισχυμένες ε, υποχρεώσεις ε, και να τις τηρεί, κάτι που δεν συμβαίνει. Ένα άλλο ερώτημα. Υπήρχαν άρθρα και στο Guardian πρόσφατα και στο παρελθόν. Είναι η εταιρεία, για την εταιρεία αυτή που σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Μάλτας προχώρησε σε μια συμφωνία ε, και έφτιαξε αυτό το σύστημα. Γνωρίζουμε πλέον ότι αυτοί είχαν σχέσεις με την Cambridge Analytica που βοήθησαν στο να τι εκλογές ε, στο Sun Kitchen Navy να κρατήσει ένα κόμμα που ήταν υπέρ αυτών των προγραμμάτων ο κύριος Αλισάνδρο ο οποίος είναι στη φυλακή στι Πολιτείε τώρα λόγω του, ε, του τραπεζικού σκανδάλου έλαβε διαβατήριο ακριβώς για να μπορέσει να ε, λειτουργήσει μια τράπεζα στη Μάλτα και τα λοιπά, έτσι. Οι Indian Partners λοιπόν είναι έτσι μια πολύ σκοτεινή οργάνωση. Σήμερα, χθες, ε, ο Guardian δημοσίευσε μία έκθεση όπου αναφέρει ότι υπήρξε lobbying προς, το, προς, το Βρετανική, κυβέρνηση για να έχουν απαλλαγή από υποχρέωση θεώρησης. Visa, visa waiver. Το ξέρω αυτό διότι την ερχόμενη εβδομάδα όλος τυχαίως έξι από αυτές τις ε, ε, δικαιοδοσίες ε, τις επικίνδυνες ε, ε, για τα προγράμματα αυτά ε, άδειας παραμονής. Ε, ετοιμαζόμαστε λοιπόν με το Μαυρίκιο, με τη Σεν Κίτσεν and με τον Μπαρμπέιντος, σε Χέλες, να υπογράψουμε Visa Waiver. Τώρα, την άλλη εβδομάδα. Καταπληκτικό, έτσι. Ε, με την ευκαιρία να πω ότι το, η, Tax 3, η Tax 3 έστειλε ένα έτοιμα προς το ε, Κοινοβούλιο πρέπει να επανεξεταστεί αυτό με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει υπό το φως του συγκεκριμένου καταλόγου. Πέρα από αυτό όμως, το ερώτημα μου είναι το εξή. Εσείς τι μάθατε για την αυτές τις οργανώσεις τις σκοτεινές, όπως οι Indian Partners, όπως η άλλη ομάδα αυτή, η οποία καλεί ε, τον κύριο Μπαρόζο ε, στα, στις του, ε, όλους αυτούς τους globalized people στους οποίους δίνουν τα προγράμματα ε, δεν βλέπουμε δηλαδή μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν βλέπουμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν λόμπι εδώ εντό θεσμικών οργάνων της Ένωσης τι εκπροσωπούν και ότι είναι κάτι ακόμα πιο σκοτεινό από ε, απλά ένα πρόγραμμα που θέλουν να βγάλουν κάποια χρήματα. Μάλιστα ευχαριστώ για το πρώτο σας ερώτημα για το θέμα της παρακολούθησης ε, στην, ε, στην ε, έκθεσή μας, στα συμπεράσματα. Δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει κάποιες τελευταίες γραμμές για, τη, για κάποιους κανόνες διαφάνειας που πρέπει να ακολουθούνται σε επίπεδο κρατών μελών. Γι' αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον αριθμό των ετούντων ανάλογα με την χώρα προέλευσης, το πόσες ε, άδειες παραμονής ε, ή άδειες ηθαγένειας δόθηκαν και πόσε δεν έγιναν δεκτές, ε, ποιοι είναι οι μεσάζοντε που εμπλέκονται στη διαδικασία και ποιο είναι ο ρόλος τους ε, ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πραγματική διαδικασία διαφάνεια σε πέντε κράτου μέλου που θα μπορούσε να συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα τώρα του ιδιωτικού τομέα, μετά την πέμπτη οδηγία, είναι ένα θέμα το οποίο το υπογραμμίζουμε στην έκθεση. Βεβαίω οι περισσότερε υποχρεώσεις αφορούν τον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε δέουσα επιμέλεια, αλλά αυτό που πραγματικά συστήνουμε εμείς στην έκθεση είναι στην περίπτωση ακριβώς των προγραμμάτων αυτών ε, η παρακολούθηση ε, από τις δημόσιε αρχές είναι εξίσου σημαντική. Και εδώ αναφερόμαστε στην ουγγρική ε, εμπειρία στην Ουγγαρία υπήρχε ένα τέτοιο πρόγραμμα ε, επενδύσεων με αντάλλαγμα ηθαγένεια και πολλές εκθέσεις έδειξαν ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή η οποία θα, ε, παρακολουθούσε την ποιότητα της διαδικασίας ε, δέους επιμέλειας, απέτυχε στο έργο της και εδώ βλέπουμε την ευθύνη των δημοσίων αρχών να εξετάσουν κατά πόσο ακολουθείται σωστά η διαδικασία δέους επιμέλειας. Τώρα για τους Indian Partners. Εδώ τίθεται πολλά ζητήματα. Ε, θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε ε, ποιο είναι το σκεπτικό όπως από την ιδέα του να υπάρχει αυτή η ιδιωτική εταιρεία η οποία ταυτόχρονα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα στο όνομα μιας κυβέρνησης, ε, κάνει το marketing αυτού του προγράμματος και οι ίδιοι είναι αυτοί που την εργούν και τη διαδικασία δέους επιμέλειας. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σε επίπεδο διαφάνεια, σε επίπεδο σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν για το ρόλο αυτών των ε, ιδιωτικών διαμεσολαβητών, μεσαζόντων. Ήσασταν στην, ε, πέρσι στην αποστολή σα, ε, εδώ αυτό προέρχεται, το βρήκαμε στην πτήση, στο αεροπλάνο τη μάλτα, όπου εδώ διαφημίζεται το πρόγραμμα, έτσι, με προσπέκτους μέσα στο αεροπλάνο. Ε, τίθεται λοιπόν πολλά ερωτηματικά, γι' αυτό λοιπόν στην έκθεσή μας εμείς συστήνουμε ε, στα κράτη-μέλη να είναι σαφή για το ποιος είναι ο ρόλος αυτών των ε, αντιπροσώπων ε, που τρέχουν το πρόγραμμα, το εφαρμόζουν και βεβαίως λαμβάνουν και χρήματα, έτσι, και αναετούντα. Ελωρίθες να προσθέσεις κάτι? πολύ γρήγορα ναι, για τις συμφωνίες ε, Visa Waiver έχει απόλυτο δίκιο. Είναι και αυτό πρόβλημα. Ε, το St. Kitts και Nevis είναι μια από τις πρώτες χώρες ε, που, έχει, που είχε πρόγραμμα CBI, έχει απαλλαγή από υποχρέωση θεώρηση με πολλά κράτη-μέλη τη Ένωση και αυτό είναι ένα στοιχείο ανησυχία που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα κράτη-μέλη ατομικά, όπω το έκανε ο Καναδά με τη Γρανάδα όταν διαφώνησαν με, με τον τρόπο με τον οποίο χορηγούν την ηθαγένεια και άλλαξαν και την πολιτική θεωρήσεων απέναντι στη χώρα αυτή. Δηλαδή μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνουν πράγματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να ζητήσω από τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον κύριο Γιάζεκ, να γράψει στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε εάν μπορούμε τουλάχιστον να καθυστερήσουμε και να επανεξετάσουμε με βάση τον κατάλογο του ΩΣΑ το συγκεκριμένη διαδικασία. Ο κύριος ε, Καντελάρη είναι εδώ. Βαντεν Καντελάρ είναι εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Ε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Όντω χαίρομαι που μπορώ να θέσω μία ερώτηση για το θέμα των χρυσών θεωρήσεων αυτών και νομίζω ότι όλοι κατανοούμε πολύ καλά τα προβλήματα και τους κινδύνους των ε, προγραμμάτων CBI και LDIs και προφανώς ε, βρωμάν, βρωμάν ε, φοροαποφυγή και διαφθορά. Από την άλλη όμως διαπιστώνουμε και τα οικονομικά πλέον και την, τον ελκυστικό χαρακτήρα τον πόλο έλξη που αποτελούν τα προγράμματα αυτά για τα κρατημέλη. Στη σελίδα 36 της μελέτης μιλάτε για τα οικονομικά ωφέλη. Και λέτε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος τέτοιων προγραμμάτων συχνά είναι πολύ αμεληταίος στην τελική ανάλυση. Ερωτώ λοιπόν, διαπιστώσατε ότι όντω πρόκειται για αμελητές ποσότητες και κατά δεύτερον αναφέρατε και εξετάσατε και ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις, ε, οι οικονομικές ε, συνέπειες, η αστάθεια που προκαλείται ως παράπλευρη απώλεια. Άρα, ποιες είναι οι, ποια είναι τα ωφέλη ποια είναι τα πλεονεκτήματα, πόσο ωφελούνται τα κρατημένα και τελικά πόσο διτεράσσεται και η οικονομία τους. Ποια είναι τα μειονεκτήματα. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική ανάλυση, λάβαμε υπόψη την άμεση εισρωή βάσει των στοιχείων που είναι δημόσια διαθέσιμα, τα οποία μας χορήγησαν οι κυβερνήσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον η ίδια επένδυση θα είχε γίνει και χωρίς το πρόγραμμα. Άρα, έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με το ύψος των επενδύσεων, δεν ξέρουμε όμως αν οι επενδύσεις αυτές θα είχαν γίνει έτσι κι αλλιώς. Σε ό,τι αφορά τώρα το spillover, τον αντίκτυπο, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί όπως σα είπαμε και πριν δεν υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει φυσική παρουσία στην επικράτεια των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τέτοια προγράμματα RBI. Δεν σημαίνει ότι θα καταστεί κανεί, για παράδειγμα, ε, φορολογητέος στην χώρα αυτή. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε πόσοι από αυτούς τους ετούντε ε, τέτοιων θεωρήσεων ζουν ή δεν ζουν στη χώρα αυτή. Άρα δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτό το αντίκτυπο, το spillover. Δηλαδή, αν ε, καταλαβαίνετε καλά τι μου λέτε, λέει ο κ. Βανδεκάντελάρα, η δυνατότητα υπολογισμού είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δεν ε, μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, εκτός και αν έχουμε κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, γιατί φυσικά το επιχείρημα που θα είχαμε κατά των θεωρήσεων θα ήταν τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση με κανέναν τρόπο. Θέλετε να απαντήσετε, λέει πρόεδρος. Εν συντομία. Κοιτάξτε, δεν είπαμε ότι είμαστε κατά οποιοδήποτε μέτρο. Απλά κάνουμε μια ανάλυση με τα αρνητικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Και όντω αποτελεί αυτό μεγάλο πρόβλημα το γεγονό ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε επαρκή στοιχεία προκειμένου να διεξαγάγουμε μια σωστή ανάλυση. Αυτό δεν είναι πόρισμα μόνο τη δική μα έρευνα, πρέπει να ξέρετε. Όχι, και το ΕΚΤ και το ΔΝΤ οι έκτη το του είχαν το ίδιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε. Η Πρόεδρος, να σας πω ότι σε χώρες όπως η δικιά μου, για παράδειγμα, η κυβέρνηση δημοσιεύει κάποια αριθμητικά στοιχεία που αποτελούν τα αποτελέσματα των επενδύσεων. Αλλά ασφαλώς οι πιο πολλές από αυτές τις χρηστές θεωρήσεις είναι για αγορές ακινήτων. Πάνω από 6.000 τέτοιες θεωρήσεις και μόνο 11 εξ αυτών χορηγήθηκαν σε άτομα που ήθελαν να ανοίξουν ε, μια επιχείρηση, μια εταιρεία που θα απασχολούσε πάνω από 10 άτομα. Και φυσικά αυτά τα στοιχεία στην Πορτογαλία συνέβαλαν πάρα πολύ στη φούσκα των ακινήτων, καθότι τα ακίνητα κατέστησαν υπερβολικά ακριβά για τους ντόπιου και έτσι τρευλώθηκε εντερός η αγορά ακινήτων σε χώρες όπως η Μάλτα όμως από την άλλη, όπου τμήμα των εσόδων των ε, διαβατηρίων και των ε, ηθαγενειών που πολλούνται πάνε στα δημόσια ταμεία, δεν υπάρχει καμία λογοδοσία για το τι γίνεται τελικά με τα λεφτά αυτά. Στη Μάλτα, για παράδειγμα, έμαθα πρόσφατα ότι τμήμα των χρημάτων που επενδύεται στο ταμείο αυτό πάει στη διάσωση ιδιωτικών τραπεζών, όπως η Τράπεζα Λαμπάρτο στην Μάλτα. Το οποίο προφανώς και είναι αξιοσημείωτο, για να το θέσουμε γενικά. Αν δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει προς τις δύο προσκεκλημένε μας, να σας ευχαριστήσουμε όλος ιδιαίτερω για την πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αυτή έρευνα και είμαι βέβαιη ότι τα πορίσματα της έκθεσής σας, της μελέτης σας θα μας αποβούν πολύ χρήσιμα. Ιδιαίτερα επειδή τέτοια προγράμματα δεν θα είχαν ε, ευδοκιμήσει αν δεν είχαν υποστηριχθεί από την Επιτροπή. Όταν ρωτάμε ερωτήσει, μα λένε Μα τι σα απασχολεί αυτό, εφόσον έχει τι ευλογίε τη Επιτροπή και στη Μάλτα και αλλού. Υποτίθεται ότι υπήρχε υποπτία και παράλληλα όλα αυτά από ό,τι φαίνεται ήταν ε, υπό τις ε, την ευλογία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα φαίνεται να ξυπνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λαμβάνει δράση. Και εμεί από πλευρά μα πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. should... Και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ δηλαδή η παρουσίαση της μελέτης που έχει θέμα του κίνδυνου νομιμοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε και φοροδιαφυγή στον τομέα των ελεύθερων λιμένων και τελωνιακών αποθηκών. Ε, στην αρχή τη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα δηλαδή, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχουμε τώρα μια μελέτη την οποία θα παρουσιάσει ο κύριος Ρόχνη, τον οποίο πολύ ορίζω, ο οποίος είναι policy analyst στο EPRS, στην Υπηρεσία Έρευνας δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και πραγματικά περιμένουμε να μας πείτε ε, τι, ε, αυτά που έχετε να, να μας πείτε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Χαίρομαι που ξανά είμαι εδώ και βλέπω τόσο οικία πρόσωπα. Τα περισσότερα τουλάχιστον είναι οικία. Τα free ports, οι ελεύθεροι λιμένες. Θα σας πω ε, στην παρουσίασή μου πρώτα απ' όλα δύο λόγια όσον αφορά τους ορισμούς. Επίσης, ε, να σας πω ότι γιατί αυξάνει τη δημοφιλία αυτών των ελευθέρων ε, λιμένων, τα προβλήματα και τους κινδύνους φόρο διαφυγής και ξεπλήματος χρήματος θα σας δώσω κάποια στοιχεία ε, νομικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια νομική ανάλυση ε, της ε, νομοθεσίας, το, την οδηγία MRB καθώς επίσης και την συνεργασία όσον αφορά τελωνιακά θέματα και φυσικά την τελωνιακή συνεργασία και τέλος θα αναφερθώ σε μια υπόθεση μελέτης και η στάτη του Freeport, του ελεύθερου λιμένα του Λουξεμβούργου. Ε, νομίζω ότι μέσα από αυτή τη μελέτη του Λουξεμβούργου μπορούμε να εξάγουμε αρκετά ε, συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία ε, ελεύθερα λιμάνια τα οποία διέπονται από τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, ένα εκ των οποίων και το Λουξεμβούργο. Ο καθορισμός των ελευθέρων ζωνών, των ελευθέρων λιμένων, καθώς επίσης και των τελωνιακών αποθηκών. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα ελεύθερα λιμάνια λιμάνια πρώτη φορά εμφανίζονται στο AMLD5, στην πέμπτη δηλαδή ε, οδηγία ε, κατά της ενομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που θα δεθεί σε ισχύ το 2020, αλλά για την ώρα δεν υφίστανται. Υπάρχει ήδη ε, δηλαδή η νομική βάση ε, για την ε, λειτουργία και την ύπαρξή τους στον τελωνιακό κώδικα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Υπάρχουν περίπου 82 free zones που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και ορισμένα είναι ελεύθερα λιμάνια. Ε, καθώς επίσης ε, και ε, τελωνιακές αποθήκες που είχαν δημιουργηθεί για τα εμπορεύματα σε διαμετακόμιση, σε τράνζιτ για την αποθήκευσή τους. Αλλά τώρα γίνονται όλο και πιο συχνά νόμιμοι βάση. Εκεί μπορεί να βρει κανείς από διαμάντια μέχρι αυτοκίνητα, μέχρι έργα τέχνης κλπ. Αργότερα στην παρουσίασή μου θα πω ότι ε, η υπάρχουν και κάποια άλλα, κάποιες άλλες αποθήκες, οι bonded warehouses, που είναι περίπου ε, σαν τις τελωνιακές αποθήκες, ε, που μπορούν να ε, παράσχουν ένα υψηλό επίπεδο αποφυγής φόρων και δασμών, που περίπου σαν τα ελεύθερα λιμάνια. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ελεύθερα λιμάνια είναι τρία, ενώ αυτού του είδους οι αποθήκες ε, είναι πολλές εκατοντάδες. Έχουμε τώρα Freeport στη Γενέβη, στο Λουξεμβούργο, στη Σιγκαπούρη, που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Μετά στο Delaware, στο Πεκίνο και άλλο ένα. Ε, είναι κοινή γνώση ότι ε, η παρουσία ενός ελεύθερου λιμανιού μπορεί να αποτελέσει ακόμα ένα σημείο έλξης και γίνεται δηλαδή το, το, το μέρος αυτό πιο ελκυστικό ως ε, Financial Center, κέντρο χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Γίνονται πολύ δημοφιλή τα ελεύθερα λιμάνια τώρα τελευταία. και δεν μπορεί κανείς να τα δει ξέχωρα από την αύξηση της δημοφιλίας ε, των έργων τέχνης ε, και της εμπορίας έργων τέχνης. Να πούμε ότι ε, ε, όλο και λιγότερο απόρριτο ε, έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις όσον αφορά το τραπεζικό απόρριτο καθώς επίσης και την φοροαποφυγή και γι' αυτό πολλοί άρχισαν να ψάχνουν εναλλακτικέ λύσεις για τα χρήματα τα οποία μπορούμε να υποψιαστούμε ότι είχαν κρύψει στις τράπεζες αυτές σε λογαριασμούς. Προσπάθησαν να βρουν αυτό που ονομάζουμε substitute assets, δηλαδή ε, ε, περιουσιακά στοιχεία υποκατάστασης, όπως ας πούμε είναι οι αντίκες ε, και, ο, και τα έργα τέχνης. Είχαμε λοιπόν μεγάλη αύξηση των έργων τέχνης και της εμπορίας τους πολύ σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι η αύξηση των μουσείων και των συλλογών τους και είχαμε μάλιστα και νέους παίκτες στην αγορά, ε, ε, παίκτες πολυεκατομμυριούχους από την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και την Ρωσία. Ε, οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν δασμούς εισαγωγής-εξαγωγής, μπορούν να, όταν στέλνουν τα, τα προϊόντα αυτά στους, στα ελεύθερα λιμάνια και επίσης οι πωλήσει, όσες φορές και αν πολιθούν τα έργα αυτά, δεν αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια για ορισμένους ανθρώπους ε, είναι ότι τα ελεύθερα λιμάνια μπορούν να δώσουν ακόμα μια διασφάλιση, ακόμα ένα επιπλέον επίπεδο ε, απορρίτου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για εμπορία και διακίνηση έργων τέχνης. Ε, ένα επιπλέον επίπεδο λοιπόν εμπιστευτικότητας και μυστικότητας προστίθεται ε, όταν περνούν τα έργα αυτά από τα ελεύθερα λιμάνια. Να πω δύο λόγια σχετικά με τους γενικούς κινδύνους όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος και την φοροαποφυγή. Ε, τα ε, ελεύθερα λιμάνια είναι εγγενώς συνδεδεμένα με την έννοια της μυστικότητας, δίνουν την δυνατότητα και επιτρέπουν συναλλαγές οι οποίες ε, ε, γίνονται χωρίς ε, να δηλωθούν ή να τραβήξουν την προσοχή των ρυθμιστών καθώς επίσης και των φορολογικών αρχών. Στις περισσότερες περιπτώσεις δηλώνει κανείς όποια αξία θέλει, όχι στο Λουξεμβούργο και επίσης κανείς δεν ελέγχει αυτήν την δηλωμένη αξία μπορεί κανείς ε, να δηλώσει μεγαλύτερη ή πολύ μικρότερη αξία. Ε, αυτό μπορεί να είναι προβληματικό βεβαίως όσον αφορά ε, και την νομοθεσία για την νομιμοποίηση παρανομών εσόδων αλλά και για τη, γενικότερα το θέμα της φοροαποφυγής. Κοιτάξτε, η επίσημη αξιολόγηση ενός ε, πίνακα, ας πούμε, μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ. Ε, και στο Λουξεμβούργο, ας πούμε, ε, μπορεί με έξοδα του Υπουργείου Πολιτισμού τα τελωνία να ζητήσουν μια αξιολόγηση του, της αξίας του πίνακα, αλλά συνήθως αυτό δεν γίνεται. Ένα άλλο στοιχείο που αφορά ακριβώς τη διεθνή αγορά τέχνης είναι ότι ε, πολλές, ε, έχει υψηλό επίπεδο ε, ε, συναλλαγών που πληρώνονται με, με μετρητά ή σε είδος. Έχουμε, ας πούμε, περίπτωση που αγοράστηκε πίνακας με 50 εκατομμύρια που πληρώθηκε με χαρτονομίσματα. Και βεβαίω ε, δεν χρειάζεται σε πολλές ε, περιπτώσεις, τι περισσότερες θα μπορούσα να πω, η φυσική παρουσία του αγοραστή. Δηλαδή ε, μπορεί κανείς να προσθέσει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης του, της μυστικότητας εάν δεν πάει ο αγοραστή στο ελεύθερο λιμάνι αλλά ένα εκπρόσωπο του όσον αφορά τον κίνδυνο φοροαποφυγής ε, ε, σε σχέση με τις ε, τελωνιακές αποθήκες. Εδώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν σε συνεργασία βάσει της DAC 5 που είναι η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία. Μερικές φορές κάποιος μπορεί μόνο να αξιολογήσει υποθετικά το, τον όγκο γιατί πολύ εν, πολύ ε, ε, πρόσφατα άρχισε να ισχύει ε, η οδηγία. Επίσης έχουμε και την πέμπτη οδηγία ε, για την ε, καταπολέμηση νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που θα τεθεί σε ισχύ το 2020. Επομένως αυτά είναι πολύ δύσκολα να μετρηθούν. Όσον αφορά τον ενωσιακό κώδικα, Αυτό θέτει μια σειρά κανόνων για την δημιουργία των τελωνιακών αποθηκών καθώς επίσης και των ελευθέρων ζωνών ή ελευθέρων λιμένων. ο UCC, αυτός ο ενωσιακός τελωνιακός ε, κώδικας, ε, επιτρέπει επίσης την ε, μη χρέωση και καταβολή έμεσων φόρων, καθώς επίσης και δασμών εισαγωγής βάσει αυτών των διαδικασιών, γιατί θεωρούνται τα αγαθά αυτά ως σε τράνζιτ, σε διαμετακόμιση. Στην ουσία επίσης οποιοδήποτε μπορεί να παρουσιάσει και να αποθηκεύσει ε, κάποιο αγαθό ε, σε μια ελεύθερη ζώνη. Ε, δηλαδή ένας δικηγόρος ή μια πινακοθήκη ή ένας έμπορος τέχνης. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στον τελικό πραγματικό ιδιοκτήτη, τον ultimate beneficial owner. Επίσης, ο τελωνιακός κώδικας ε, ε, θέλει να ε, πιάσει και την έμεση φορολόγηση και επομένως ενδιαφέρεται για το ίδιο το αγαθό και όχι τόσο πολύ για τον ιδιοκτήτη. Όσον αφορά τα τελωνία, ε, πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ και ο δασμός και δεν τον ενδιαφέρει απαραίτητα ε, ε, ποιος είναι ο τελικός, ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Ε, τώρα, κάποια συμπεράσματα. Ο τελωνιακός κώδικας ε, δίνει ε, μια νομική βάση για την αποφυγή των έμεσων φόρων και επίσης δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης σε τελωνιακές αποθήκες μέσα από ειδικέ διαδικασίες αποθήκευσης εάν τα αγαθά αυτά διακινούνται και πολλούνται ή αγοράζονται εντός του ελευθέρου λιμένος, ε, τότε οπωσδήποτε δεν έχουν καταβληθεί οι έμεση φόροι. Όπως είπα και προηγουμένως, ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να αναφέρω στα συμπεράσματα είναι ότι σχεδόν οποιοδήποτε μπορεί να ε, φέρει σε μια τελωνιακή αποθήκη ή σε ένα ελεύθερο λιμάνι ε, οποιοδήποτε αγαθό και ο πραγματικός ιδιοκτήτης μπορεί να βρίσκεται μίλια μακριά. Και επίσης ε, μπορεί ο ε, ε, ιδιοκτήτης να ζητήσει αποθήκευση υπό το ίδιο καθεστώς αλλά σε μια άλλη αποθήκη που μπορεί να έχει ας πούμε στην, στις Βρυξέλλες και όχι απαραίτητα στο ελεύθερο λιμάνι. Προχωράω τώρα ε, στο θέμα της νομοθεσίας κατά της νομοποίησης παρανόμων εσόδων. Ε, όπως σας είπα, επανειλημμένα θα τεθεί σε ισχύ τη 10η Ιανουαρίου του 2020 ε, και εκεί θα, αναφέρεται, ε, θα αναφέρονται και τα ελεύθερα λιμάνια καθώς επίσης και στις αρχές και τους οικονομικούς ε, φορείς που μπορεί να είναι πινακοθήκες, που μπορεί να είναι ε, δημοπρατικές ε, εταιρείες κλπ. Αυτά, αυτές οι εταιρείες θα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. Οπωσδήποτε προβλέπεται και η καταχώρηση όλων των θεωρούμενων υπόπτων ε, συναλλαγών. Όσον αφορά τώρα την τέταρτη γενιά της AML, ε, αυτή τέθηκε σε ισχύ τη 10η Ιουνίου του 2017 και έχει προσθέσει τα tax crimes, ε, δηλαδή φορολογικές παράνομες πράξεις, οι οποίες μπορούν και οφείλουν να καταγράφονται. Είναι γεγονός ότι υπάρχει αύξηση ε, των καταγγελιών ο αλλά στο Λουξεμβούργο ας πούμε ανεπίσημα έμαθα ότι έχουν περίπου 600 ε, δηλωμένες ε, ως ύποπτες κινήσεις από τον Ιούνιο του 2017. Επίσης, ε, οι αρχές ε, οι οποίες ασχολούνται με την άμεση φορολογία θα έχουν πρόσβαση μετά από αίτημα, upon request, ε, στα στοιχεία τα οποία βασίζονται στην δέουσα επιμέλεια που με τη σειρά τους βασίζονται στην πέμπτη οδηγία για την διοικητική συνεργασία. Σας δίνω εδώ ένα μικρό σχέδιο. Of ε, θέλησα λίγο να μελετήσω το κατά πόσον οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες και αν και κατά πόσον ε, είναι ανταλλάξιμες, αν υπάρχει δηλαδή ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών ιδεοδός από το 2020 οι αδειοδοτημένοι ε, οικονομικοί παράγοντες των ελεύθερων λιμένων θα πρέπει να δίνουν πληροφορίες και για τα προϊόντα αλλά και για την ταυτοποίηση του ε, ε, ιδιοκτήτη οι πληροφορίες ε, για τον Ultimate Beneficial Owner ε, θα πρέπει να ε, δίνονται στην εποπτική αρχή. Και αυτό μετά από αίτημα βάσει της DAC 5. Θα δίνονται οι πληροφορίες λοιπόν στο ε, στην υπηρεσία των άμεσων φόρων, αλλά δεν θα είναι ένα απλό αίτημα δώσ' μου όλα τα στοιχεία ας πούμε, που έχεις. Θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη ε, υποψία, έτσι ώστε να δοθούν στοιχεία για τον τελικό ιδιοκτήτη. Ε, και βεβαίως αυτό είναι ε, ε, κατά κάποιο τρόπο αφαιρεί νόημα από την διαστασιμότητα με την έννοια ότι δεν μπορείς να έχεις βάσιμες υποψίες από τη στιγμή που δεν ξέρεις τι αποθηκεύεται ε, σε αυτές τις αποθήκες. Ίσως τα πράγματα αλλάξουν σε σχέση με το 2000, μετά το 2020 γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ζητηθούν και δεν είναι καθόλου προσβάσιμες οι πληροφορίες για τον τελικό πραγματικό χρήστη. Επίσης δεν υπάρχουν ακόμα οι αρχές επιτήρησης AML. Και επομένως η μόνη πληροφόρηση που μπορεί να υπάρχει είναι από τους αδειοδοτημένους ε, ε, operators. Για το MLD θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Κάτι που πιστεύω το AMLD5. Μία παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δεν συνάδει η ορολογία που χρησιμοποιείται στο MLD με τον ε, τρονιακό κώδικα. Για παράδειγμα, οι ελεύθεροι λιμένες, ε, οι οποίοι θεωρούνται ε, ως μία οποιαδήποτε άλλη ελεύθερη ζώνη. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει είναι κατά πόσον ε, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή το MLD5 σε εφαρμογή θα συμπεριλαμβάνει και τις αποθήκες για παράδειγμα. Αυτό θα έχει τεράστια, τεράστιες επιπτώσεις. Για το κατά πόσον θα συμπεριληφθούν οι αποθήκες με το αντίστοιχο επίπεδο Όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν πρωτού τεθεί σε εφαρμογή. Η νομοθεσία EU AML βασίζεται στην καλή πίστη και στην εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων οντοτήτων, όχι σε συστημικές ανταλλαγές που θα απαιτούσαν αυτόματη διαβίβαση στοιχείων. Δεν υπάρχουν συστημικές λοιπόν τέτοιες ανταλλαγές πληροφοριών των στοιχείων αυτών AML. Η μελλοντική επιτυχία του AMLD, της οδηγίας κατά της ε, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πηγές, εξαρτάται από τον υψηλό βαθμό αποτρεπτικού παράγοντα σε ό,τι αφορά, ό,τι αφορά τη μελλοντική εποπτεία, καθώς και στην ε, δίωξη για την επιβολή κυρώσεων. Ξέρουμε πώς πήγαν τα πράγματα στον τραπεζικό κλάδο και καλό θα ήταν να το κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα αυτό πριν από το 2020. Και τώρα να περάσω στην οδηγία για την διοικητική συνεργασία, DAC, DAC. Η DAC 1, η πρώτη τέτοια οδηγία, προβλέπει αυτόματη ανταλλαγή μεταξύ των ε, φορολογικών υπηρεσιών, ε, προκαθορισμένων δεδομένων φορολογικής φύσης, σε τακτική φύση, στην βάση σε ό,τι αφορά τους υπηκόους σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η πρώτη τέτοια οδηγία λοιπόν προβλέπει ανταλλαγή κατόπιν ετήματος και ευθελούσιες ανταλλαγές μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η γενική διατύπωση. Και όπως σας είπα, η πέμπτη τροποποίηση της οδηγίας, η DAC 5, δίνει τη δυνατότητα στις ε, φορολογικές υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση με κατόπιν ε, αιτήματος σε πληροφορίες UBO που συλλέγονται από AML. Και εδώ να προβούμε σε κάποια συμπεράσματα και κάποια πορίσματα να δούμε. Όταν πολύ κανείς ένα πίνακα σε έναν ελεύθερο λιμένα τον αγοράζει 5 εκατομμύρια, τον πουλάει 2 εκατομμύρια, ε, 7 εκατομμύρια, συγγνώμη, 2 εκατομμύρια κέρδο, κεφαλαϊκό κέρδο, το οποίο όμω δεν είναι το ίδιο σε κάθε χώρα. Ενδεχομένω λοιπόν να χρειαστεί να το αναφέρει ο πολιτής είτε όχι. Είναι κάπως θεά αυτή η ζώνη σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών, τέτοιες πωλήσει και ε, κεφαλαϊκά κέρδη δεν υπάγονται στο DAC 1, στην πρώτη τέτοια οδηγία. Οι αποθήκες και πάλι υπάγονται στην οδηγία κατά το ξεπλήματο χρήματο, στην AMLD, γιατί αυτό θα έδινε πρόσβαση στις υπηρεσίες σε τέτοιες πληροφορίες σε όλες αυτές τις αποθήκες και μιλάμε για χιλιάδες στον αριθμό. Επίσης, οι φορολογικές υπηρεσίες ε, δεν ε, μπορούν να έχουν τέτοια πρόσβαση σε δεδομένα UBO. Έχουν πρόσβαση κατόπιν ετήματος μόνο. Αυτό στην πράξη δυσκολεύει, δυσχεραίνει πάρα πολύ την πρόσβαση, γιατί είναι χρονοβόρα διαδικασία. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν κάποιος αντίκτυπος όταν υπάρχει κάποια υποψία και μπορεί να υποβάλει έτοιμα στα εμπλεκόμενα μέρη ή μπορεί να λάβουν πληροφορίες από φορολογικές υπηρεσίες άλλου κράτους μέλους. Αλλά πραγματικά συστημικά ωφέλη δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Δύο λόγια τώρα για το Λουξεμβούργο να πω. Ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί έχει βάλει τον ελεύθερο λιμένα του στο καθεστώς ε, της οδηγίας νομιμοποίησης ε, παρανόμων εσόδων το 2015. Προσαρμόστηκαν λοιπόν και πήραν ε, και την άδεια τη σχετική προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή για την οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματο και άρα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση να δούμε κατά πόσο είναι επιτυχημένη η οδηγία η MLD5 και είναι μοναδική περίπτωση υπό την έννοια ότι έχει μόνιμο αποδεκτικό χώρο ε, διαφορετικών πολύτιμων αγαθών στα πλαίσια του λιμένα της Γενεβής. Οι εμπλεκόμενοι φορείς στο Λουξεμβούργο, όπως ε, σας είπα, στο μέσα βλέπετε, στη μέση του διαγράμματος βλέπετε τους ε, εγκεκριμένου ε, διαχειριστές ελεύθερων πάνω τις ε, υπηρεσίες έμεσης φορολόγησης και τον επόπτη AML κάτω τα τελωνία που είναι υπευθυνή για τα προϊόντα και για τους έμεσους φόρους, αριστερά το, της FIU, της Εθνικές Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικών Μονάδων και στα δεξιά τις ε, παρολογικές υπηρεσίες για τον άμεσο φόρο. Αν και στην περίπτωση του Λουξεμβούργου αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη πρακτική εφαρμογή. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε πώς ε, γίνεται η αναφορά ύποπτων συναλλαγών στο Λουξεμβούργο. Κάθε αρχή θα πρέπει να αναφέρει προς το, τη μονάδα οικονομικού κινδύνου. Από τη Δελωνία, η υπεύθυνη με την οποία συνομίλησα μας είπε ότι υπήρχε αναφορά 4-5 φορές προς ε, την μονάδα αυτή. Έγινε μια αναφορά σε έναν Έλληνα υπηκό στη λίστα Λαγκάρντ. Υπήρχαν υποψίες κατά αυτού, αλλά και υποψίες σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια τα οποία παρουσιάστηκαν η, έμεση, η ομάδα έμεσου φόρου είναι στο Λουξεμβούργο και ο υπευθύνο ΕΠΟΠ της AML. Άρα, το 2015 τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία AML. Ε, δόθηκε μία περίοδος χάριτος ενός έτους για να ασκηθεί η τέουσα επιμέλεια, να γίνουν σχετικέ έρευνες, να ενημερωθούν τα δεδομένα και στη συνέχεια ξεκίνησε ο έλεγχο, ο διασταυρούμενο έλεγχο, κατά πόσο πραγματικά υπήρχαν σωστά, σωστή τήρηση δεδομένων και έτσι έλαβαν έναν κατάλογο δεδομένων από τα τελωνία και με τον κατάλογο αυτό ελέγχθηκε διασταυρούμενα με τους ε, παρόχους κατά πόσο να όλα αυτά. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Σε τις περιπτώσεις μάλλον που δεν υπήρχε η συμμόρφωση αυτή, έγινε αναφορά στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι διαχειριστέ των αδειών μας είπαν ότι έχασαν 30 περίπου πελάτες ε, του ετέθησε σε εφαρμογή η οδηγία AML. Προφανώς δεν τους άρεσε η ιδέα ότι θα αποκαλύπτουν τα ταυτότητά τους στις σχετικές αρχές. Επίσης ε, έχουν αναφερθεί μια σειρά από υποψίες προς τους FIUs από αυτούς που διαχειρίζονται τις άδειε. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν αναφορές, είναι βεβαίως ε, μοναδικό αυτό στον τομέα των ελεύθερων λιμανιών. Τώρα το θέμα της ε, διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και του και τη διαμήραση των πληροφοριών. Το εξήγησα και νωρίτερα. Θα δείτε εδώ πιο κάτω ότι έχω βάλει κάποιες γραμμές με ε, διακεκομένα, διακεκομένες γραμμές ε, όταν είναι κατόπιν ετήματος, περιορισμένη δηλαδή η πρόσβαση εδώ. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα ανταλλαγή στα πλαίσια του ΦΑΤΚ ε, που έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια του ΩΣΑ ή την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία. Ε, αυτή η δυνατότητα είναι κατά τη γνώμη μου έτσι πολύ περιορισμένη. Επίσης έχω βάλει διακεκομένη γραμμή διότι αυτός που διαχειρίζεται την άδεια ε, στο Λουξεμβούργο μου επιβεβαίωσε ποτέ δεν ζητήθηκε πληροφορία από την αρμόδια αρχή. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, είμαι αρκετά βέβαιος ότι δεν έχει λάβει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών του Λουξεμβούργου και των συναδέλφων τους σε άλλες χώρες. Και τώρα έρχομαι στις τελευταίες ε, ε, ε διαφάνειες στα συμπεράσματα για το Λουξεμβούργο. Οι αρχές επικεντρώθηκαν ε, κυρίως την έμεση φορολόγηση που σχετίζεται με αποθηκευμένα αγαθά και όχι σε φόρο ή ενδεχόμενη επίπτωση στο φόρο εισοδήματος. Οι διαδικασίες τηλωνιακές του Λουξεμβούργου είναι εξαιρετικά αυστηρές όλα ελέγχονται. Οι αξιωματικοί εκπαιδεύονται από τους ειδικού του, του Υπουργείου Πολιτισμού να μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους πίνακες, να γνωρίζουν κατά πόσο κάποια έργα τέχνης είναι πλαστά ή ε, υπερτιμημένα. Ε, τα τελωνία λοιπόν έχουν πληροφορίες για τα δεδομένα, αλλά για τα αγαθά μάλλον, αλλά χρειάζονται τη νομική βάση για να το μοιράζονται ε, με άλλες αρχές, ε, όπως με τι φορολογικέ αρχέ, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τι επιπτώσει στο φόρο εισοδήματο λόγω των κεφαλιακών κερδών μετά από την πώληση ενό εργοτέχνης, το τελωνίο ενημερώνεται για το νέο ε, ιδιοκτήτη αν δηλαδή συστηματικά κάτι που πολίτες σαν ελεύθερο λιμάνι να ε, ενημερώνουν για την πώληση αυτή οι φορολογικές αρχές, ε, θα είχαμε άμεσε επιπτώσεις. Ε, θα είχαμε άμεσο αντίκτυπο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει νομική βάση και δεν υπάρχει τέτοια νομική βάση στο Λουξεμβούργο. Είναι το μόνο ελεύθερο λιμάνι ε, υπό το καθεστώ AML στον κόσμο. Βεβαίω εξαρτάται από την πειθαρχία που επιδεικνύουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο είναι στεγανό. Η πρόσβαση στις πληροφορίες τώρα από ε, την φορολογική, την, τις υπηρεσίες άμεσης φορολόγησης, ε, εδώ είναι δύσκολο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει πρόσβαση, είναι και το πιο σημαντικό σημείο συμπερασματά μου. Αυτά. Ευχαριστώ, Ρον, πραγματικά συναρπαστικά αυτά που ακούσαμε. Ε, βρήκατε πολλά στοιχεία, όλη τη δυσκολία ε, το πόσο συχνά ε, πόσο συχνά είναι οι πηγές ε, θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις παρακαλώ ο κ. Βαντεκάντελάρε Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε για τον και για τον κόσμο των ελευθέρων λιμανιών και για τον κόσμο του εμπορίου έργων τέχνης. Ε, αναφερθήκατε κάποια στιγμή στο γεγονός ότι οι αποθήκες δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο. Ε, το λογικό ερώτημα λοιπόν είναι ποιος ε, θα μπορούσε να είναι κατά να συμπεριληφθούν οι αποθήκες στους κανόνες αυτούς. Δεν υπάρχει κάποιο λογικό επιχείρημα γιατί να μην συμπεριληφθούν οι αποθήκε, ιδιαίτερα αν δει κανεί τα στοιχεία, τα αριθμητικά. Επίση, ε, αν συγκρίνουμε ε, ελεύθερε ζώνε σε τρίτε χώρε, όπω στη Σιγκαπούρη, στη Γενέβη, ε, τα, ε, τα, τα ελεύθερα λιμάνια στην Ευρώπη φαίνεται να ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίω, άλλο τι λέει θεωρία και άλλο τι λέει πράξη και άλλο τι γίνεται στην πράξη, αλλά τα ερωτήματα είναι ε, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι περαιτέρω ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα αλλάξει τον τρόπο ή μάλλον θα, θα διώξει τους ανθρώπους αυτούς από τα ευρωπαϊκά ε, ασφαλή λιμάνια ε, οπότε θα χάσουμε κάθε έλεγχο δηλαδή έχει νόημα να συνεχίζουμε να νομοθετούμε ταυτόχρονα όμως ρωτάω υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω νομοθεσία εφόσον είναι στα χέρια, στα των κρατών μελών να, να σεβαστούν αυτή την νομοθεσία ή όχι. Παραδείγματο χάρη υποχρέωση αναφοράς το αν σέβονται, γίνει σεβαστά αυτό ή όχι, ε, δεν είναι κάτι που ούτε καν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Υπάρχουν δηλαδή δύο όψεις του δύο νομίσματος στην πραγματικότητα. Είναι ενδιαφέρον αυτό με τα ελεύθερα λιμάνια, αλλά αφενός ε, θέλουμε να διώξουμε κι άλλο ε, και να χάσουμε έλεγχο, να διώξουμε αυτούς που το χρησιμοποιούν με νέα νομοθεσία, ε, η οποία όμως ε, θα έχει και κενά ή θα μεγαλώνει κενά που ήδη υπάρχουν. Ε, μπορεί να μου απαντήσετε σε αυτό το δίλημα. Με το πρώτο ερώτημά σας πρώτα για τις αποθήκες που πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο της οδηγίας μπορεί να μην είναι σαφή δεν είναι 100% σαφέ κατά πόσο συμπεριλαμβάνονται ή όχι. Το, η διατύπωση στο, OM, το OMD5 ε, είναι αντικείμενο διαφόρων ερμηνεών. Εγώ πιστεύω ότι βεβαίω θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι αποθήκε ε, στην ίδια νομική βάση με αυτή του τελωνιακού κώδικα ο, ε, όσο ό,τι δηλαδή ισχύει για τις ελεύθερες ζώνες θα πρέπει να ισχύει και για τι αποθήκε. Τώρα, κατά πόσο είναι πρόβλημα αυτό, ποιο θα έχει πρόβλημα με αυτό. Ακούστε, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποθήκες για ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται, μετακομίζουν, χωρίζουν και αυτές οι αποθήκες μπορούν να ζητήσουν άδεια για να αποθηκευσούν και αποθηκευτούν εκεί αγαθά που βρίσκονται σε τράνζιτ. Συνήθως υπάρχει κάποιος σε ένα γραφείο εκεί, ε, τίποτα δεν ελέγχεται, βεβαίως δηλώνονται τα αγαθά αυτά στο τελωνίο, Αλλά για να υπάρξει πραγματική ιδέουσα επιμέλεια, ε, για να, για να δηλαδή, γίνουν σεβαστέ οι σχετικέ απαιτήσει, θα πρέπει να γίνουν τεράστιε προσπάθειε από, από του ε, διαχειριστέ αυτών των αποθηκών. Ε, δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό δηλαδή. Από την άλλη, αν αν, εφόσον δεν ρυθμίζονται οι αποθήκε και ρυθμίζονται τα ελεύθερα λιμάνια, θα, θα δούμε αυτό που συμβαίνει και στην Ελβετία πριν η Ελβετία γίνει μέλος του Παγκόσμιου Οργάνωσης Εμπορίου, είχε πολλά ελεύθερα λιμάνια και στη συνέχεια, μετά την ένταξη στον ΠΟΕ, ε, δόθηκε η δυνατότητα να υπάρχουν και αποθήκες τελωνιακές και οι κανόνες ήταν πολύ πιο χαλαροί εκεί από ό,τι στα ελεύθερα λιμάνια. Πριν πολλά ελεύθερα λιμάνια έκλεισαν στην Ελβετία και αυξήθηκαν οι αποθήκες το ελεύθερο λιμάνι της Γενέβης βεβαίως πάντα ήταν ε, εξαιρετικά ελκυστικό διότι είναι το κλασικό μέρος όπου μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει ένα πίνακα του Πικάσο. Σχετίζεται αυτό και με την, ε, το Art Fair της Βασιλείας. Ε, εάν πάντως δεν ρυθμίσει κανείς ε, τις αποθήκες, είναι, πολύ εύκολα θα πάρουν τη θέση των ελευθερών λιμανιών. Εγώ στο ελεύθερο λιμάνι θα ζήταγα άδεια να αλλάξω καθεστώ και να γίνω αποθήκη τελωνιακή. Τώρα για τη Σιγκαπούρη, τη Γενέβη ε, και ναι, στο Λουξεμβούργο ρυθμίζεται πολύ περισσότερα πράγματα από ότι εκεί. Είναι αυστηροί οι κανόνε τελωνιακοί και υπάρχει και το EML. Μπορεί να, αμφισβητήσει κάποιο την αποτελεσματικότητα του EML βέβαια, αλλά υπάρχει το σύστημα για την καταπολέμηση του συλλογικού χρήματο. Στη Γενέβη υπήρξαν επικρίσεις από τους ε, επίσημους ε, κρατικούς ελεγκτές. Έκτοτε ε, άρχισαν να εισαγάγουν ένα, μια κάποια δέουσα επιμέλεια, αλλά δεν, δεν έχουν φτάσει να υποχρεώσουν ε, τις ε, διάφορες επιχειρήσεις να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη των αγαθών. Αυτό που βλέπετε λοιπόν στο Delaware, στο Μονακό, στο Hong Κόνγκ, στο Πεκίνο, ε, στη Γενέβη υπάρχει ένα ανταγωνισμό του πόση ουσιαστικά μύθια προσφέρει ο καθένας. Καλό είναι να γνωρίζουμε, παραδείγματο χάρη, είναι ο κ. Μπουβιέ, ο ιδιοκτήτη του Λουξεμβούργου, είναι και ο μεγαλύτερο μέτοχο του, ε, του ελεύθερου λιμανιού στη Γενέβη και έχει και άδεια να επιχειρήσει. Στη Γενέβη είναι και έμπορος τέχνης, είναι και στη Σιγκαπούρη, είναι και σύμβουλος στο Πεκίνο και έχει μπλέξει σε αρκετά σκάνδαλα. Οι αρχές του Λουξεμβούργου βαλένουν δεν είναι έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι το σκάνδαλο στο οποίο έχει μπλέξει σχετίζεται και με την εισαγωγή του AML για την, ε, το ελεύθερο λιμάνι του Λουξεμβούργου. Ε, είναι προφανώς ε, μία δουλειά η οποία έχει μια μυστικότητα και υπάρχει μια ανταγωνισμός για το πώς η μυστικότητα μπορεί να προσφέρει το κάθε ελεύθερο λιμάνι. Τώρα για την αγορά έργων τέχνης ε, είναι ενδιαφέρον αυτό. βεβαίως δεν έφτασα στο σημείο να μπορώ να αναφερθώ στον αντίκτυπο στην αγορά έργων τέχνης στην Ευρώπη ε, αλλά σίγουρα θα υπάρξει αντίκτυπο ε, ε, εφόσον μπορούμε να ξέρουμε ποιο ποιος πουλάει το έργο αν είναι μια εταιρεία που ανοίξει μια άλλη εταιρεία και αυτή με τη σειρά σε μια άλλη εταιρεία, ε, θα πρέπει τότε να τεθούν ερωτήσεις. Ε, ξέρετε, η μυστικότητα σε αυτή τη δουλειά, σε αυτόν τον κόσμο, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν ρωτάει κανεί, δεν πρέπει να ρωτάει κανείς. Και είναι εύκολο βέβαια κάποιο να μετατοπίσει την εταιρεία του εκτό Ευρώπη. Μπορεί να υπάρξουν λοιπόν τέτοιου ε, επιπτώσει. Τώρα, ε, ακόμα και αν έχουν όλε τι πληροφορίε για του δικαιούχου και του ιδιοκτήτε οι αρχέ, ε, οι φορολογικέ αρχέ έχουν πρόσβαση μόνο κατόπιν αιτήματο. Πρέπει να υπάρχει ήδη μια υποψία εκ των προτέρων για να έχει κάποιο πρόσβαση στι πληροφορίε αυτέ. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα οι επιπτώσει δεν είναι και τόσο μεγάλε για τους δικαιούχους. Δηλαδή μπορούν να περάσουν κάτω από το ραντάρι αν θέλετε. Ακόμα και έτσι και με αυτή την, ε, την εφαρμογή. Τι μπορεί να γίνει για τη μελλοντική νομοθεσία, είπατε. Είναι σημαντικό καταρχήν να υπάρξει να ευθυγραμμιστεί, το MLD με τον τελωνιακό κώδικα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε να κάνετε κάτι για τον κίνδυνο ξελπάνους χρήματος σε ελεύθερα λιμάνια, ένας τρόπος είναι το AML, αλλά και ένας άλλος είναι ο τελανιακός κώδικας. Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να περιορίσουμε την διάρκεια που μπορεί να μείνουν σε τράνζιτ τα έργα Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του πλανιακού κώδικα. Κάτι άλλο. τα ε, έργα τέχνης ε, ε, είναι περιζήτητα για τους επενδυτές. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και καλύτερη ρύθμιση της αγοράς έργων τέχνης, να υπάρχει κάποιος επενδυτικός τίτλος και ο οποίος να ρυθμίζεται για τα έργα τέχνης. Ελπίζω να απαντώ στα ερωτήματά σας. Πίτερ. Καταρχάς, ε, μια παρατηρήση, επιτρέψτε μου. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι πολλοί από τους ομιλητές ε, δεν είναι παρόντες και θα είχαμε κανονικά 25 Ομιλητέ, μήπω να καλέσουμε τον κύριο Τόμας να έρθει λίγο πιο νωρίς για το επόμενο θέμα, για να μην παραταθεί περαιτέρω αυτή η κατάσταση, γιατί νομίζω ότι δεν ε, επιδεικνύει τον απαραίτητο σεβασμό αυτό προς το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να περάσουμε και στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Ρωτώ λοιπόν. Ε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και όσο πιο πολύ σας ακούω, τόσο πιο πολλά ερωτήματα γίνονται στο μυαλό μου και σε εσά ε, φαντάζομαι. Αν κάποια στιγμή λοιπόν αποδεχτεί αν υποθέσουμε ότι όλοι τηρούσαν το EML και να δούμε τι γίνεται στο Λουξεμβούργο. Έχουμε έναν νοικιαστή ο οποίος αποθηκεύει προϊόντα. Θα πρέπει να αποδείξει ποιος είναι ο, οικονομικά, ο, ο, ιδιοκτήτης, ο οικονομικός ιδιοκτήτης. Και αν αυτός ο, ο ιδιοκτήτης πουλήσει περαιτέρω σε κάποιον άλλον τα προϊόντα αυτά, πώς θα βεβαιωθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα καταλήξουν στον ε, ενοικιαστή και στη συνέχεια και στην υπηρεσία στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ε, Μήπως έτσι ανοίγουμε πάλι το κουτί της Πανδώρας, μήπως ο ενοικιαστή μπορεί να πει πάλι ότι δεν το γνώριζε. Κατά δεύτερον, αναρωτιέμαι το εξή. Σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο σύστημα, πώς ε, θέλετε να επιβληθούν κυρώσεις και ήταν αυτό είναι από τα θέματα που θίξατε. Αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές, ε, υπάρχει σε ποινικό επίπεδο, δεν υπάρχει κάτι ευρωπαϊκό, ούτε σε ό,τι αφορά τη δημόσια τάξη. Τι εργαλεία θα είχαμε λοιπόν στην διάθεσή μας για να στραφούμε κατά ενός κράτος μέλους ή να υποχρεώσουμε ένα κράτος ε, να προβλέψει τέτοιες κυρώσεις όταν δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να παρέμβουμε. Και μία τρίτη ερώτηση τουλάχιστον για τώρα, γιατί έχω πάρα πολλές ερωτήσεις ακόμα. Ποιος θα ελέγξει τελικά τι αποθηκεύεται. Να δούμε για παράδειγμα τα αυτοκίνητα. Έχω ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα. Εδώ τα πράγματα είναι μάλλον απλά. Μπορεί να ελεγχθεί βάσει των δεδομένων καταχώρησης ποιο αυτοκίνητο είναι. Σε ό,τι αφορά τα ε, έργα τέχνης, τα πράγματα δυσκολεύουν σε αντίκες. Είναι σχεδόν αδύνατον να υπάρξει διασταύρωση στοιχείων. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει ε, αστυνομική έρευνα, για παράδειγμα, η οποία ποτέ δεν θα τελεσφορήσει και ε, δεν μπορεί κανείς να κοιτάει όλες ε, τις αποθήκες και να βρει τι, ότι υπάρχει ένα άγαλμα αρχαιολενικό με χαρακτηρισμό Αφροδίτη, Δίας. Πώς θα ελέγχουν οι φορολογικές αρχές ότι όντως στην αποθήκη περιλαμβάνεται το προϊόν το οποίο αναφέρεται. Είναι τόσες πολλές οι δυνατότητε που υπάρχουν σε σχέση με την αποθήκευση προϊόντων. Και αυτό χωρίς να λάβουμε υπόψη τον κίνδυνο φοροδιαφυγής ε, και απάτης. Μήπως απλά δημιουργούμε τις τέλειες συνθήκες για κάθε εγκληματία στην Ευρώπη. Η Πρόεδρος, πρώτο απαντήσατε να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Και στη συνέχεια θα ζητήσω από τον Πίτερ να με αντικαταστήσει, γιατί θα πρέπει δυστυχώς να φύγω. Αλλά σίγουρα θα ενημερωθώ για την απάντησή σα. Αυτά που είπατε με βρίσκουν σύμφωνοι. Συνάδουν και με αυτά που είδαμε όταν ε, επισκεφθήκαμε το ελεύθερο λιμένα του Λουξεμβουργού. Εδώ στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά και τις απαντήσεις που λάβαμε από τις αρχές ε, του Λουξεμβούργου πριν από την ημέρα πριν από την ε, ομιλία του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου στην Ολομέλεια. Όντως, ε, αδιαφάνεια, μυστικότητα και στη συνέχεια έλεγχη υποτυπώδης. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταρτίζουμε νομοθεσίας. Το θέμα όμως πάντα είναι η υλοποίηση, η συμμόρφωση και η έλεγχη, η σοβαρή έλεγχη. Και αυτή είναι ανυπαρκτή, γιατί όλα αυτά έχουν φτιαχτεί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των εγκληματικών οργανώσεων, των ε, κυκλωμάτων ξεπλήματος χρήματος αναφερθήκατε στον κόσμο της τέχνης. Δεν είναι μόνο το θέμα τα έργα τέχνης και αυτοκίνητα και διαμάντια, χρυσός. Και εικονικές εταιρείε. Προφανώς ε, όσο αποδεχόμαστε το σύστημα των εικονικών τέτοιων εταιριών. Ε, μπορεί κάνει να τις αποθηκεύει εκεί. ως ε, πρωθυπουργός, ως ε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις εικονικές αυτές ε, εταιρείε. Το σουηδικό, το ελβετικό μοντέλο, συγγνώμη, έχει να κάνει με τη Γενέβη. Δεν πιστεύετε ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να κάνει μια έρευνα στα όλα λιμένα της Γενέβης για να διασφαλίσει ότι και εκεί θα υπάρξουν ε, επιπτώσεις, όχι μόνο για τα κρατη που έχουν ελεύθερους λιμένες όπως το Λουξεμβούργο ή αποθηκευτικούς χώρους με παρόμοια συστήματα. Η Γενέβη, ωστόσο, και η Ελβετία φέρει ιδιαίτερη ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές ε, τις ερωτήσεις. Στη Γενέβη έχουμε περίπου αποθηκευμένες ε, 1,2 ε, εκατομμύρια εργατέχνες ε, που η αξία τους ξεπερνάει τα 100 δις ε, ελβετικά φράγκα. η σύγκριση με την η σύγκριση Γενέβης και Λουξεμβούργου ε, θα πρέπει να είμαστε ας πούμε στο Λουξεμβούργο πολύ ε, σαφείς σχετικά με τα εισαγόμενα ε, γνωρίζουν τι εισάγεται και την αξία τους στην Ελβετία, από ό,τι μαθαίνω, anything goes, οτιδήποτε μπορεί να μπει ε, δηλαδή μπορεί να δηλώσει κανείς ότι ε, βάζει έναν πίνακα αξίας 100.000 ευρώ και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να δώσει καμία άλλη ε, διευκρίνηση. Όπως και με τα Panama Papers δημιουργήθηκαν εταιρείε για να αποφύγουν φόρους και τα λοιπά. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα παράνομο. Ε, γίνεται παράνομο από τη στιγμή που δεν δηλώνονται ε, τα ε, στοιχεία στις φορολογικές αρχές και που δεν γίνεται γνωστή η ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ε, ε, δεκάδες ε, καλοί λόγοι για να διαλέξει κανείς το Λουξεμβούργο. Δηλαδή, η ασφάλεια, μια και μιλάμε για προϊόντα τέχνης, για έργα τέχνης, οι καλές συνθήκες όσον αφορά την υγρασία κτλ. Ξέρετε ότι η ασφάλεια και το, ο τρόπος συντήρησης των έργων τέχνης, επειδή μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, είναι κάτι το οποίο λαμβάνουν υπόψη ε, οι ενεχόμενοι κυρώσεις όσον αφορά την μη αναφορά non-reporting. Κοιτάξτε, η φοροαποφυγή, ε, η φοροδιαφυγή είναι οπωσδήποτε παράνομη πράξη ε, βάσει του, ε, μη, ε, του, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της του ξεπλήματος χρήματος, αλλά εδώ μιλάμε για εταιρείες οι οποίες δεν θεωρούνται και επομένως δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ε, ε, πινακοθήκες ή μπορεί να είναι γκαλερί τέχνης ή μπορεί να είναι ε, δικηγόροι ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ε, απλά. Δεν είναι τράπεζες οι τράπεζες οι οποίες ε, υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα έχουν λύσει αυτά. Όσον αφορά το τι γίνεται όταν ο beneficial owner, ο τελικός, ο πραγματικός ιδιοκτήτης πουλήσει το έργο τέχνης. Μα αυτό σημαίνει Ε, ότι μπορεί το έργο τέχνης να μετακινηθεί από τη μία πλευρά της αποθήκης σε μια άλλη, ενώ η πραγματική χρηματική συναλλαγή να λάβει χώρα στην άλλη πλευρά του κόσμου. Και ε, ούτως ή άλλως οι τράπεζες πλέον είναι υποχρεωμένες να ε, κάνουν την αναφορά. Και επαναλαμβάνω ότι η πραγματική μεταφορά μπορεί να γίνει οπουδήποτε και η οικονομική μεταφορά επίσης μπορεί να γίνει οπουδήποτε και μπορεί κανείς να επιλέξει κάποιο σύστημα που να μην είναι τόσο διαφανές. Ähm, Τέλεια. Ο κύριος Κόμπερν είναι στον κατάλογο και χαιρόμουν που θα πάρει το λόγο για να συζητήσουμε. Αλλά θα τον βλέπω στην αθούσα. Ο κύριος Νίτερ Μάιερ, ο οποίος και αυτός δεν είναι παρόν, ο κύριος Κάντελάρα, ούτε αυτός είναι και η κυρία Άννα Γκόμες, ούτε αυτή είναι εδώ και άρα να παρακαλέσω τον μοναδικό συνάδελφο στην αίθουσα μήπως έχει να κάνει καμία ερώτηση μετά από όλα αυτά τα απίστευτα που ακούσαμε και είναι πραγματικά κρίμα, κρίμα που δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι να ασχοληθούν εντελεχώς με τα θέματα αυτά, με ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε ζητήσει, συζητήσει. Στις επιτροπές, γιατί το θέμα του ξεπλήματος χρήματος των διεθνών επιχειρήσεων με τα Panama Papers, όλα αυτά μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν. Αλλά το θέμα των ελεύθερων λιμένων έχει χιλιάδες αδευκρίνηστες ερωτήσεις. Χιλιάδες ερωτηματικά για το πώς μπορούμε καν να το επιλύσουμε το θέμα αυτό στην Ευρώπη. και θα έπρεπε να δώσουμε το μήνυμα από τη δική μας Επιτροπή ότι έχει έρθει η στιγμή να αντιδράσουμε. Ίσως είναι άτυχη η σημερινή χρονική στιγμή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα παρά το γεγονός ότι η ώρα είναι μόλις 4 ε, και 10 να περάσουμε στο τρίτο πανέλ και να κοιτάξουμε τις εταιρείε ε, γραμματοκιβωτίων και να ακούσουμε την κυρία Ιβάνα Κνικρίστλ, αναλυτρία πολιτικής, ε, για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της, ε, τα αποτελέσματα της έρευνας, της έρευνας σας και τη συνεργασία της με την κυρία Τύριον. Thank you, Chair. And thank you for the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας εδώ για τις εταιρείες προπετάσματα, όπως τις λέμε, shell companies. Το επόμενο τέταρτο λοιπόν θα μιλήσω καταρχήν για τον όρο Shell, οι εικονικές εταιρείες, δηλαδή τι εννοούμε ακριβώς όταν μιλάμε για Shell Company. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως αυτή η η, η έννοια βεβαίως όσο ξέρετε καλύτερα από όλους τα τελευταία χρόνια αλλά δεν αναφέρεται πάντα στο ίδιο πράγμα. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς τώρα. Θα εντοπίσουμε τρεις βασικούς τύπους ε, shell companies, εικονικών εταιριών και θα εξηγήσουμε ε, τον κάθε τύπο. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για δεδομένα ε, ή για την έλλειψη καλύτερα δεδομένων ε, για τις Shell Companies και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τους δείκτες. Ε, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, αναζητήσαμε ε, δείκτες οι ενδείξεις για την ύπαρξη αυτών των εικονικών εταιριών. Και εκεί έχουμε διάφορους τύπους δικτών και θα τους εξηγήσουμε. Η συνάδελφος Χελοντή στη συνέχεια θα μιλήσει για τους διάφορους κινδύνους που συνδέονται με τους τρεις τύπους ε, εικονικών εταιριών και τον αντίκτυπο. Επίσης η Ελλοντή θα μιλήσει και για τις ε, υπάρχουσες πολιτικές ε, καθώς και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές για να μπορέσει να μετριαστεί ο κίνδυνος, οι κίνδυνοι που απορρέουν από την ύπαρξη αυτών των εταιριών. Λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι ήταν μια καλή ιδέα ε, να πούμε πρώτα απ' όλα για το τι δεν είναι αυτή η μελέτη. Δεν είναι ένα case study του Shell Company. Δεν λέμε ακριβώς τι αποτελεί Shell Company. Δεν περιλαμβάνουμε εδώ τα trust, τα ιδρύματα και άλλες, άλλες, άλλες περιφερειακές δομές και στο γεωγραφικό ε, πεδίο δεν καλύπτουμε τα υπερπόντια ε, διαμερίσματα και τα προπόνια εδάφη της Ένωση. Μιλάμε για το έδαφο τη Ευρωπαϊκή, Ένωση όπως το ξέρουμε, δηλαδή στην Ευρώπη. Λοιπόν, κάποιου όρου καταρχήν. Ε, χρησιμοποιείται συχνά ο όρο εικονική εταιρεία, Shell Company. Όμως ε, συχνά ε, τον το ανταλλάσσουμε με άλλους όρου. Letterbox Company, ταχυδρομική θερίδα, δηλαδή, ε, εντότητες ειδικού σκοπού κτλ. Αυτοί οι όροι όμως δεν αναφέρονται πάντα στο ίδιο πράγμα. Ε, κάναμε μία μελέτη της βιβλιογραφίας και διαπιστώσαμε ότι ε, ανάλογα με το πλαίσιο ορίζονται διαφορετικά ε, αυτέ, αυτές οι εταιρείε. Και με βάση λοιπόν το πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται έχουμε δημιουργήσει τρεις τύπους εικονικών εταιρεών. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ ένα νέο ορισμό, έτσι, ε, αλλά θέλουμε να περιγράψουμε για ποιο πράγμα μιλάμε ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται. θα δούμε πρώτα θα δούμε λοιπόν αυτούς τους τρεις τύπους ε, shell companies. Μιλάμε για ανώνυμες εικονικές εταιρείε, ταχυδρομικές θηρίδες και οντότητες ειδικού σκοπού. Εδώ τα βλέπετε. Οι ανώνυμες ε, εικονικές εταιρείε, ε, προφανώς το βασικό στοιχείο εδώ είναι η ανωνυμία, ο τελικός δηλαδή δικαιούχος, ο ιδιοκτήτης κρύβεται ε, μέσω διαφόρων διακανονισμών ε, πίσω και εδώ μιλάμε βεβαίως για διαφθορά, φοροδιαφυγή, εξέφλημα χρήματος ε, και χρηματοδότηση τρομοκρατικών ε, ενεργειών κτλ. Ε, εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις, αλλά καλό είναι να το διαχωρίζουμε. Ο δεύτερος τύπος είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς ε, Letterbox Company, μια εταιρεία ταχυδρομική θηρίδα, δηλαδή μια εταιρεία που είναι, καταγεγραμμένη είναι καταγεγραμμένη σε ένα κράτος μέλος, με μια οικονομική δραστηριότητα όμως που λαμβάνει η χώρα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτές οι εταιρείε συχνά χρησιμοποιούνται για να μπορέσει κάποιος να ε, ε, παρακάμψει εργατική νομοθεσία, εθνικούς κανόνες, ε, προσπάθειες δηλαδή παράκαμψη συνήθως της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και η τρίτη κατηγορία είναι αυτές οι οντότητες ειδικού σκοπού σημαντικές ε, οντότητες, ε, μιλάμε συνήθως για πολυεθνικές εταιρείες, ε, το χρηματοδότηση ομίλων, holding, τα έχουμε συμπεριλάβει εδώ, διότι συχνά γίνεται αναφορά σε αυτές σε ό,τι αφορά την φοροαποφυγή και τον επιθετικό φορολογικό προγραμματισμό ας πούμε. Είδαμε λοιπόν αυτές τους τρεις τύπους εικονικών εταιριών και εξετάσαμε τώρα, το εξετάσαμε από το πρίσμα της ε, επιτροπής σας, δηλαδή έχοντας κατά νου το δικό σας ενδιαφέρον. Αν μας είχε ζητηθεί, παραδείγματος χάρη, να παρουσιάσουμε ε, τις εταιρείε αυτές ε, στην Επιτροπή Αποσχόλησης, δεν θα μιλούσαμε ε, για την για το Letterbox Company. Αν ήταν, ήταν να μιλήσουμε στην Επιτροπή ITER, θα επικεντρωνόμασταν στις ανώνυμες εταιρείε. Ε, δηλαδή, πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Ε, δεν είναι αυτή μια κατηγοριοποίηση πάντως καιρού των εικονικών εταιριών, ανάλογα με το που εστιάζει κάθε επιτροπή, προσαρμοστήκαμε και εμείς. Τώρα που διευκρινίζαμε λοιπόν για ποιο πράγμα μιλάμε, ε, όταν λέμε για εικονικές εταιρείε, shell companies, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στα δεδομένα αυτών των ε, εταιριών. Είναι λίγα τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν πλήρη αξιόπιστα στοιχεία για τις εικονικές εταιρείε. Ιδιαίτερα για τους δύο πρώτους τύπους. Δηλαδή τους τύπους. Λοιπόν, τα πράγματα είναι καλύτερα σε ό,τι αφορά τις οντότητες ειδικού σκοπού. Εκεί έχουμε στοιχεία, συνδέονται και με τις άμεσες εξωτερικές επενδύσεις, ε, οπότε εκεί έχουμε αρκετές, ε, αρκετά στοιχεία από αξιόπιστες πηγές. Αυτή η έλλειψη δεδομένων ε, που αφορά όλους τους τύπους εικονικών εταιριών ε, μας οδήγησε στο να ακολουθήσουμε μια έμεση προσέγγιση και να αναζητήσουμε δείκτες Ενδείξει παρουσίας τέτοιων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ το σκεπτικό μας ήταν απλό. Έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στα πλαίσια των προηγούμενων επιτροπών ε, και των διαφόρων leaks ε, ότι συχνά ο αριθμός των εταιριών αυτών ε, σχετίζεται με μια σειρά από χαρακτηριστικά. Εξετάσαμε λοιπόν μια σειρά από χαρακτηριστικά που συνδέονται με την παρουσία των εικονικών εταιριών, επιλέξαμε τρία χαρακτηριστικά ε, που είναι οι καλύτεροι δείκτες, ας πούμε, οι καλύτερες ενδείξεις για να έχουμε μια εικόνα για την ύπαρξη των εικονικών εταιριών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι τα εξή. Ε, που ανήκουν σε, σε σε ένα κράτος μέλος το ποσοστό των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ ενός κράτους μέλους και επίσης το κενό κέρδους ανάμεσα στις ε, ε, εταιρείε ε, τις εγχώριες και τις εξωτερικές σε ένα κράτος μέλος. Ε, να σας πω τώρα τι βρήκαμε. Αυτός είναι ο πρώτος δείκτης πόσες εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς βρίσκονται στο κράτος μέλος. Ε, εδώ πρέπει να πω καταρχήν κάτι που έχει σημασία. Ε, μπορεί να είναι προφανές, αλλά καλό είναι να το τονίσουμε. Όλες οι εικονικές εταιρείες ανήκουν ε, σε αλλοδαπούς, αλλά όλες οι εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς δεν είναι απαραίτητα και εικονικές εταιρείες. Έτσι, εν πάση το έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσοστό ξένων εταιριών ε, ως δείκτης. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σαφές εδώ ε, στην οθόνη σας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφώς ο πιο δημοφιλής, ο πιο προορισμός, αν θέλετε, και ακολουθείται από τρεις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και μετά έχετε η Γαλλία Εστονία, Ρουμανία και Σλοβακία και μετά η Γαλλία. Αυτά είναι τα στοιχεία, εκτιμήσεις βέβαια είναι αυτές. Πρέπει να έχουμε κατά νου όμως και το μέγεθος της χώρας. Η Εστονία, παραδείγματο χάρη, μια χώρα 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει περίπου τον ίδιο αριθμό ξένων εταιριών με τη Γαλλία. Ε, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Για το πρώτο δίκτυο, λοιπόν, συνοψίζοντα, ο αριθμό των εταιριών που ανήκουν σε ξένου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο, σαφώ, μετά οι τρει χώρε τη Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και μετά η Γαλλία. Η μελέτη στην οποία βασιστήκαμε ε, δεν έδινε στοιχεία αναχώρα για τις υπόλοιπες 75.000 εταιρείες αυτός είναι ο αριθμό ο οποίος διαιρείται μεταξύ των 23 κρατών μελών. Και τώρα περνάμε στον δεύτερο δείκτη. Είναι οι άμεσες εξωτερικέ επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εδώ αυτό δεν το πήραμε σε απόλυτου αριθμούς, αλλά ως ποσοστό για να λάβουμε υπόψη μα και το μέγεθο τη κάθε χώρα. Και εδώ τα ευρήματα όπως βλέπετε στην οθόνη δεν, βλέπει κανείς και πολλά πράγματα σε αυτό το, αυτό το διάγραμμα. Το πρώτο κράτος μέλος πολύ ψηλά σε σχέση με τους άλλους είναι το Λουξεμβούργο όπου έχουμε ε, μεγάλα αποθέματα πάνω από 57 του ΑΕΠ, στοιχεία από το 2017. Αυτά το ποσοστό για άλλες χώρες ε, μπορεί να μοιάζει πολύ πιο χαμηλό, αλλά αν το δούμε λίγο πιο κοντά, διαπιστώνουμε ότι και πάλι ε, είναι πολλαπλάσια του ΑΕΠ της χώρας. Ε, στη Μάλτα, παραδείγματος χάρη, 17 φορές το ΑΕΠ, έτσι, το εσωτερικ, οι εσωτερικές ε, ε, άμεσες εξωτερικές επενδύσεις ε, και οι εξωτερικές 7 φορές. Ε, στην Κύπρο είναι 900 φορές το ΑΕΠ, ε, στην Ολλανδία 535, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία πάνω από 300%, ε, υψηλά ποσοστά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις άμεσες εξωτερικές επενδύσεις σε σχέση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Γιατί έχουμε λάβει πόσο στο στοιχείο αυτό διότι δίνεται εδώ στο έμφαση στο ποσοστό ε, από ό,τι φαίνεται ένα μεγάλο μέρος αυτών που είδατε στις προηγούμενες πίνακες ένα μεγάλο μέρος των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων βρίσκονται στα χέρια των ε, οντοτήτων ειδικού σκοπού. Ε, βεβαίως ε, αυτό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι κυρίως το τελευταίο σημείο εδώ, γιατί λέει πολλά αυτή η διαφάνεια. Αυτές οι οντότητες ε, ειδικού σκοπού δεν δημιουργεί πραγματικές επενδύσεις σε μια χώρα είναι οικονομικές ροές που περνούν από τη χώρα αυτή. Μεταφέρονται δηλαδή ροές από μη κατοίκους της χώρας προς άλλους μη κατοίκους της χώρας. Δηλαδή μπορεί να μοιάζει με επένδυση ένα κράτος μέλος. Μπορεί το πρώτο κομμάτι δηλαδή της ροής να φτάνει στην χώρα αυτή, αλλά μετά φεύγει. Τέλος, ένα υψηλό ποσοστό των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων ε, ε, αφορά τις οντότητε ειδικού σκοπού. Αυτό βλέπουμε σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, πάλι στο Λουξεμβούργο πάνω από 90% και προς τα έξω και προς τα εσωτερικό σε ό,τι αφορά τι άμεσε εξωτερικέ επενδύσει. Ε, αφορούν δηλαδή ε, τι οντότητε ειδικού σκοπού. Το ίδιο ισχύει για, το, για, τη Μάλτα και για τι κάτω χώρες Συνοψίζοντας τον δεύτερο αυτό δίκτυ, οι άμεσες εξωτερικές επενδύσεις, αν συγκρίνουμε με το ΑΕΠ της κάθε χώρας και το ποσοστό των δοτήρων ειδικού σκοπού σε αυτή τη εξωτερική επενδύσει, όλα αυτά μα δείχνουν ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν πολύ υψηλέ ε, εξωτερικές άμεσες επενδύσεις και εδώ αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2017 και, τις, και τις σχετικά ευρήματα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, να εξηγηθεί μερικώς μόνο από πραγματική οικονομική δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στο ίδιο το κράτος μέλος. Επιπλέον η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και οι κάτω χώρε έχουν υψηλό ποσοστό των άμεσων εξωτερικών επενδύσεων ε, που ε, είναι στα χέρια των ρωτήτων ειδικού σκοπού. Αυτά για το δεύτερο κριτήριο. Αυτός ήταν ο δεύτερος δείκτης και εδώ έχουμε το τρίτο και τελευταίο. Ε, είναι η διάσταση ε, αποδοτικότητας μεταξύ ξένων και ε, γηγενών ημιδαπών εταιριών στα κράτη-μέλη. Εδώ βλέπουμε ε, μεγάλη διαφορά, μεγάλη διάσταση στην Ιρλανδία, στο Λουξεμβούργο και μετά κάτω χώρες και Βέλγιο. Δεν θα πω τίποτα άλλο πέρα από αυτούς τους τρεις ε, δείκτες ε, και θα δώσω το λόγο στην Ελλοντή για να σας μιλήσει για αξιολόγηση κινδύνου ε, όσον αφορά αυτές τις ίδιες εταιρείες αλλά ε, και τους κινδύνους ε, τους γενικότερα που απορρέουν από αυτές. Θα ήθελα από το πρώτο τμήμα της παρέμβασης να διατηρήσετε ότι υπάρχουν τριών ειδών εικονικές εταιρείε. Έχουμε λίγα στοιχεία όσον αφορά ε, κυρίως τις δύο πρώτες μορφές και τέλος ότι κανένας από αυτούς τους τρεις δείκτες που ανέφερα προηγουμένως δεν αποτελούν απόλυτα, ε, απόλυτα στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης ε, των εταιριών αλλά οι δείκτες ε, συνδυασμένες και με άλλα συγκυριακά στοιχεία ε, καταδεικνύουν την ύπαρξη των εικονικών εταιριών σε διαφορετικό βαθμό και βαρύτητα στις διάφορες χώρες μέλη. Ελοντή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω εγώ τόσο πολύ. Θα σας παρουσιάσω τους κινδύνους ε, που σχετίζονται με την κακή χρήση των shell companies πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσουμε ότι οι shell companies ε, μπορεί να έχουν ε, νομιμοποιημένους ε, σκοπούς και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε joint venture και ειδικού σχεδιασμού κινήσεις και από μόνες τους δεν αποτελούν κίνδυνο. Ωστόσο, όταν σχετίζονται, σχεδιάζονται με την ανωνυμία και με τους αποσπασμένους εργαζόμενους μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν με εσφαλμένο τρόπο. Ε, έλεγα ότι αυτές οι shell companies, λαμβάνοντας υπόψη και σε συνδυασμό με στοιχεία τα οποία ανέφερε η Σνάτσο προηγουμένως, δίνουν την δυνατότητα ανωνυμία ε, στους ε, ε, ιδιοκτήτες, ενώ έχουν την δυνατότητα οι ιδιοκτήτες αυτοί να χρησιμοποιήσουν για όποιο λόγο θέλουν την εταιρεία και ανεφέρθηκε προηγουμένως τρομοκρατία, διαφθορά κλπ. Αυτού του είδους ε, η εικονική ε, εταιρεία ονομάστηκε Anonymous Shell Company, ανώνυμη εικονική εταιρεία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εταιρείε αυτές έτσι ώστε να παρακαμφθούν ε, και να καταπατηθούν διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες. Μέσω λοιπόν μιας τέτοιας shell company δίνεται η δυνατότητα ε, να ε, ε, χρησιμοποιηθεί μια τρίτη οδός μέσω της οποίας δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που βάσει συμβάσεων απορρέουν και θα έπρεπε να εφαρμοστούν στις σχέσεις μεταξύ δύο χωρών. Ε, αυτές είναι κυρίως οι special purpose entities, δηλαδή οι οντότητες ειδικού σκοπού. Ε, μέσω τέτοιου είδους εταιριών μπορεί κανείς ε, να κορφολογήσει την πιο απλή διαδικασία όσον αφορά ε, τις εργασιακές συνθήκες κλπ. Τρίτος λόγος χρήσης αυτών των εταιριών είναι η αποφυγή των κοινωνικών διατάξεων που σχετίζονται με την εργασία των εργαζομένων. Επιλέγεται δηλαδή αυτή η μορφή εταιρείας έτσι ώστε να αποσπώνται εργαζόμενοι αποκλειστικά ε, από χώρα με υψηλά κοινωνικά, υψηλές κοινωνικές εισφορές σε άλλη χώρα με χαμηλές κοινωνικές εισφορές. Ε, κυρίως σε αυτή την κατηγορία ε, εμπίπτουν οι letterbox companies. Προφανώς τέτοιες εσφαλμένες χρήσεις των shell companies έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο μπορεί να αποτελέσουν ε, ε, εστίες ε, δυνητικού, δυνητικών διαδικασιών ξεπλήματος χρήματος, φόρο αποφυγής, φόρο διαφυγής, τρομοκρατίας, διαφθοράς κλπ. Μπορεί να έχουν αντίκτυπο γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία, ας πούμε μέσω αρνητικής επίπτωσης στο ΑΕΠ, ανάπτυξη παρανόμων εγκληματικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων, ε, μείωση της εμπιστοσύνης ε, στους θεσμούς κλπ. Εάν ε, θέλουμε να, τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να μειώσουν την, τον αντίκτυπο αυτών των εταιριών, λαμβάνουν διάφορα, διάφορα μέτρα, όπως ας πούμε η πλήρης απαγόρευση Shell Company στη Λετωνία. Υπάρχουν ενδιάμεσες εταιρείε οι οποίες πλέον δεν έχουν την δυνατότητα ε, να ε, έχουν σχέσεις με shell companies. Το καλοκαίρι στην Λετωνία ο αναπληρωτής κυβερνήτης Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι ε, η το ξεκαθάρισμα των, ε, ε, της οικονομικής εικόνας της χώρας ε, από αυτές τις shell companies είχε έναν αντίκτυπο της τάξης μόνο του 0,5% ε, στο ΑΕΠ, ωστόσο για να έχουμε τον πραγματικό αντίτυπο, αντίκτυπο θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν συμφωνεί με τόσο δραστικές ε, προσεγγίσεις. Αντιθέτως θα θεωρεί ότι είναι καλύτερα η αντιμετώπιση κάθε μίας από τις τρεις μορφές εταιρείας. Πρώτα απ' όλα βάσει της οδηγίας κατά του του ξεπλήματος ε, παράνομου χρήματος. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις Shell Companies, αναφέρει ότι ε, όλες οι εταιρείες ε, οι οποίες εμπίπτουν στην ε, κατηγορία της άρσης της ανωνυμίας στο τέταρτο και πέμπτο δίκτυο AML, άρα και οι Shell Companies, θα πρέπει να εφαρμόζουν και να υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες. Δεύτερον, πολλά μέτρα προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά την παράκαμψη των ε, συνθήκων. Ε, ας πούμε, μέσω της Parent Subsidiary Directive, επίσης και μέσω της τροποποίησης της ε, βάσης, της φορολογικής ε, ε, βάσης και της μεταφοράς των κερδών. Υπάρχουν επίσης και άλλα τρία νομοθετήματα τα οποία οπωσδήποτε θα μειώσουν όταν εφαρμοστούν τον κίνδυνο που απορρέει από τις οντότητες ειδικού σκοπού και τις ανώνυμες εταιρείες. Πρόκειται ε, για, τις, ε, για το CBCR καθώς επίσης και το CCTB και το CCCTB. Γίνεται μια προσπάθεια διασύνδεσης ανάμεσα στην φορολόγηση ε, και την χώρα στην οποία παράγεται το κέρδος και με τον τρόπο αυτό οπωσδήποτε η επίπτωση στις Shell Companies θα είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, ε, ε, η Enforcement Directive καθώς επίσης και η αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους και την απόσπαση εργαζομένων μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά την δυνατότητα των letterbox companies να παρακάμπτουν τις συνθήκες. Τέλος, Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα περισσότερα μέτρα μετρίασης, μετριασμού συγγνώμη, ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρόσφατα μέτρα. Επιπροσθέτως, ε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση πολλά νομοθετήματα. Επομένως, είναι πάρα πολύ νωρίς ε, για να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιδράσει αυτή η ισχύουσα νομοθεσία και η μελλοντική νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να δούμε και την ε, διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών ε, ε, πράξεων ε, σε σχέση με αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, χρυσές θεωρήσεις και ελεύθερα λιμάνια. Θα πρέπει να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να δούμε πόσο, και πόσο καλά, με ποιο τρόπο και πόσο καλά λειτουργούν όλα αυτά τα διοικητικά μέτρα. Ευχαριστώ. Και η διοικητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και για τη δουλειά που κάνατε για μας. Πρώτος, ε, στο μετάλλαγο των ομιλητών, ο κύριος Τόμας Μάννα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα που μιλάει και ο πρόεδρος. Ναι, μα μιλάω τόση ώρα γερμανικά. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Τάξη 3 θεωρώ ότι είχαμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με την επικεφαλή της ομάδας κώδικα διοντολογίας και εγώ και εμ, κάποιοι συνάδελφοι αμφισβητήσαμε τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων μόνο εφόσον ε, ε, τέθησε την προοπτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαφανίστηκαν 9 ε, από τις 17 αυτές χώρες ε, από τον κατάλογο αυτό, ως διαμαγείας. Και έτσι λοιπόν αυτές οι απειλές φαίνεται ότι έχουν αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα φορολογικά συστήματα τα οποία έχουν κατάλογα, κατά χαρακτήρα προδιαφυγής και είναι πολύ εξελιγμένα αυτή η ανάγκη ανώνυμία σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσει, επιχειρήσεις, όλες οι καταχρήσει που αναφέρατε και η οδηγία για τους αποσπασμένους που για μένα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό θεωρώ να φροντίσουμε κάπως να καταπολεμήσουμε την ε, το παράνομο αυτό το χρήμα στην Επιτροπή Ταξένα και Ταξιδία και στην Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά. Εξετάσαμε το πού θα πρέπει να καταβάλλονται οι φόροι, εκεί που είναι το κέρδος, εκεί που δημιουργείται η θέση απασχόλησης και να μην δημιουργούνται διαρκώς εικονικές ε, επιχειρήσεις. Όταν η επιλογή ενός, ε, μιας έδρας ε, έχει να κάνει με τους φόρους που α, μπορεί να γλιτώσει κανείς. Γιατί συχνά το θέμα είναι ότι ακόμα τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για τους φόρους. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα την οποία θα επιθυμούσαμε. Το Justice Network ε, δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα που καλεί για ανάληψη δράση, γιατί υπάρχουν τέσσερα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην κορυφή των ranking που ε, αποσχεπούν τέτοια στοιχεία για φοροδιαφυγή. Τι μέτρα λοιπόν μπορούν να λεφθούν για να αποτρέψουμε τέτοιες ε, πρακτικές βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και τι μηχανισμούς έχετε να προτείνετε. Γιατί να λέμε απλά ότι υπάρχουν εικονικές επιχειρήσεις ε, τις οποίες θέλουμε να καταπολεμήσουμε, αλλά να μην έχουμε νομικά εργαλεία δεν αρκεί. Και επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουμε λάβει ως μέτρα ως τώρα. Γιατί υπάρχουν διαρκώς τέτοιες απόπειρε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε Περιορισμένε ευθύνε, αλλά πάντα έχουμε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που έχουμε και αν θα μπορούσαν οι πολίτες να διαβάσουν αυτά που έχουμε πετύχει, θα καταλάβαιναν πόσο σημαντικά είναι. Γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν φόρου ζωή να διατηρούνται, ότι είναι δική του η αρμοδιότητα. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να το κοιτάξουμε αυτό στον προεκλογικό αγώνα από όλα τα πολιτικά κόμματα, αγαπητέ Πρόεδρε για να δούμε τι είναι δίκαιο, γιατί θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αδικία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και προς ποιον θέσατε την ερώτησή σας, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Και πράγματι η κατάσταση όπως διαγράφεται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο μάτι του κυκλώνα. Έχει περάσει τόσο μεγάλος όγκος νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια. Νομοθεσία η οποία πρόσφατα μόνο έχει τεθεί σε εφαρμογή και ενδεχομένω θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον, που είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, δεδομένης δε και ε, του χαρακτήρα διαπλοκής ε, του προβλήματος. Η νομοθεσία λοιπόν υφίσταται και αναφέρατε σημαντικές νομοθεσίες οι οποίες θα έπρεπε να εγκριθούν. Και μετά από κάποια χρόνια μόνο θα διαπιστώσουμε ποιος είναι ο αντίκτυπος και πώς ε, γίνεται η υλοποίηση, αν υπάρχει πραγματική εφαρμογή ή όχι. Και αν επιτυχάνονται τα αποτελέσματα που είχαμε υπόψη μας. Η εφαρμογή λοιπόν θα είναι κρίσιμος παράγοντας. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, νομοθεσίας η οποία εύκολα υπονομεύθηκε στην βίβλο του 2015 η οδηγία για τις, ε, για τα, τις οικονομίες, για τους λογαριασμούς στην Ελβετία που ανήκουν σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε η οδηγία για τις, ε, τα ποσά αυτά ετέθησε σε εφαρμογή και αποτέλεσε τεράστιο πρόβλημα αυτό ότι τεράστιο ποσοστό των λογαριασμών δεν είναι και πλέον σε φυσικά πρόσωπα αλλά μεταφέρθηκε στην ιδιοκτησία ε, επιχειρήσεων, εταιριών. Αυτό προέκυψε λοιπόν από τις μελέτες μας ότι υπάρχει σαφής ε, α, σχέση με τον αριθμό των εταιριών. Δεν μπορούμε όμως να διακρίνουμε τι άλλα παραθυράκια υπάρχουν γιατί στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΟΝΤΗ αναφέρθηκε στη διασύνδεση διάφορων νομοθετημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θεωρούμε ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχετε μήπως κάποια ερώτηση προς τον κύριο Μαν. Ναι, στην ε, περώτηση ξέρετε ότι οι ευρωβουλευτές ε, που θέλουν να πετύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Τι θα μας εστήνετε λοιπόν να κάνουμε για να ξεκαθαρίσουμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να υπάρξει μετατόπιση των αρμοδιοτήτων σε φορολογικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να πούμε, να λέμε συνέχεια. Σας παρακαλώ αγαπητό Συμβούλιο, αξιοθείτε να εξετάσετε το αίτημά μας πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση. Υπάρχουν ε, δημοσιογράφοι, ερευνητές οι οποίοι μας βοηθούν, αλλά ενδεχομένως να μην υπάρχει αυτό. Εσείς τι θα συστήνατε. Ζητώ συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό μας βασανίζει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει νομοθετική αρμοδιότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ασκήσουμε πολιτική πίεση. Πιστεύω δε ότι οι συνάδελφοι εδώ ενδεχομένως να μην ε, ε, έχουν εμπειρία σε ό,τι αφορά την πολιτική πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε εμείς, η πολιτική, αλλά αν υπάρχει κάποια νομοθετική δυνατότητα να ασκηθεί πίεση, θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Αλλά η τροποποίηση των συνθήκων και η άσκηση πολιτικής πίεσης είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων. Θα είμαι σύντομη. Με την νομοθεσία που συμφωνήθηκε και πάλι χρειάζεται μια αξιολόγηση, αλλά σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση των εικονικοτεριών στην Ευρώπη, χωρίς να είμαι επερισιόδεξη, φαίνεται ότι πλέον έχει δρομολογηθεί η νομοθεσία και η νομοθεσία θα αποτρέψει τις καταχρήσεις τέτοιων εικονικών εταιριών. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο τύπο που διαπιστώνουμε στην αναθεώρηση. Το θέμα είναι βασικά η εφαρμογή, αλλά ενδεχομένω τα απορίσματα της Επιτροπής απασχόληση να έχουν πιο πολύ σημασία στο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το τρίτο σκέλος, τα τεράστια ποσά που ρέουν εισραίουν προς τις εντότητες ειδικού σκοπού, σε ό,τι αφορά και τα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα κάποιων χωρών, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξη, φαντάζομαι τη επιτροπή Τάξ 2 και τη Τάξ 3. Θα πρέπει να δοθούν λοιπόν συγκεκριμένες συστάσεις γιατί οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ΑΣΑ θα μπορέσουν μόνο από κοινού να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ελπίζω να σας ικανοποιεί αυτό ως απάντηση. Σας ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος. Επόμενος από το ΕΛΚ. Είμαι εγώ και έχω μία ερώτηση να κάνω σε ό,τι αφορά την κλειδονία την οποία αναφέρατε. Μας ε, δείξατε με πολύ καλό τρόπο τι δείκτες υπάρχουν για να εντοπίσουμε τις εικονικές εταιρείε. Η Λετωνία αν απαγορεύσει ολοσχερός ε, τις ε, εικονικές εταιρείε θα πρέπει να έχουν κάποιες ε, ορισμούς για το τι αποτελεί εικονική εταιρεία. Όταν κάνει κανείς το χύψη, θεωρείται εικονική εταιρεία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, ποιε είναι αυτέ οι προδιαγραφέ και μήπω θα μπορούσε αυτό να μα οδηγήσει ή να δώσει μια ένδειξη για μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή λύση. Η απάντηση. Από τεχνικής άποψης δεν απαγορεύτηκαν οι εικονικές εταιρείε. Απαγορεύτηκαν οι εμπορικές ε, σχέσεις με τις εικονικές αυτές επιχειρήσεις. Ναι, αλλά και γι' αυτό χρειάζεται ο ορισμός, λέει ο πρόεδρος. Ο ορισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι στη σελίδα 33 της ε, έρευνας. Αν θέλετε να ρίξετε μία ματιά εκ παραλληλού. Οι εικονικές λοιπόν αυτές εταιρείε δεν έχουν σύνδεση νομικού προσώπου με οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή ή ε, δράση οικονομικού προσώπου με μηδαμινή άμα, οικονομική αξία και δεν υπάρχει οποιαδήποτε τεκμήριο που θα αποδείκνει το αντίθετο. Οι κανόνες και η νομοθεσία της χώρας όπου είναι καταχωρισμένη η εταιρεία δεν προβλέπουν υποχρέωση αναφοράς οικονομικών δραστηριοτήτων στις οικονομικές μονάδες του εκάστοτε κράτους, όπως είναι οι αιτήσεις λογαριασμοί και το νομικό πρόσωπο δεν έχει χώρο ή για άσκηση οικονομικών δράσεων στην ε, χώρα όπου ρεύει η εταιρεία. Εναλλακτικά οπου εδρεύει η σωρευτικά, σωραστικά λεει ο Πρόεδρος. or. Είναι διαζευτικό το e. Ist aus Ihrer Πιστεύετε ότι αυτά που εξετάσαμε στη Λετωνία είχαν αποτέλεσμα. Μπορούμε να αποδείξουμε κατά πόσον μειώθηκαν, για παράδειγμα, οι αλλοδαπές επενδύσεις στην Λετωνία μετά την εισαγωγή της νομοθεσίας. Τον Απρίλιο εγκρίθηκε ο νόμος. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να σας πούμε τι έγινε ακριβώς, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε τους δείκτες που σας παρουσιάσαμε, γιατί οι πιο πολλοί διεκτέ ήταν του 2015. Άρα του χρόνου θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκόπιμο και πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε τα ίδια οικονομικά στοιχεία και να δούμε πραγματικά ποιο ήταν ο πραγματικό αντίκτυπο. Τελευταία ερώτηση από πλευρά μου, λέει ο πρόεδρο, σε ό,τι αφορά του κατόχου τέτοιων εικονικών εταιριών. Που συχνά χρησιμοποιούν ε, ξύπνους ε, οικονομικούς διαχειριστές, ε, και αφήνουν την οργάνωση της όλης κατάστασης ε, στα έμπειρα χέρια τέτοιων διευθυντών. Σε ό,τι αφορά τη Λετωνία, στην μελέτη σας ε, έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο καλύτερης ε, διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εταιριών αυτών που αναλαμβάνουν την οργάνωση τέτοιων εικονικών επιχειρήσεων. Ähm, Και δεν μιλάω μόνο για χρηματοοικονομικές υπηρεσίε. Συχνά πρόκειται για δικηγορικά γραφεία, μεγάλε εταιρείε συμβουλευτική ε, Τράπεζα ενδεχομένω. Αλλά μήπω ε, έχετε κάποια στοιχεία για το πώ αυτοί οι εταίροι που υποστηρίζουν το στήσιμο μιας εικονική επιχείρηση, μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που θα θεσπιστεί. Δηλαδή έχει ως στόχο κυρίως τους μεσάζοντες. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξή. Έχετε δώσει σημεία αναφοράς. Έχετε να πείτε ότι κοιτάξτε εδώ και εκεί πρέπει να κινηθούμε παραπέρα γιατί αυτό δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη και ως Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Στην έκθεση μας επικεντρωθήκαμε στους τρεις τύπους εικονικών εταιριών στις οποίες αναφερθήκαμε και στην ανάλυση μας έως τώρα οι περισσότερες ανησυχίες αντιμετωπίζονται με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία ή με την νομοθεσία που βρίσκεται από προπαρασκευή. Θα πρέπει να γίνει πρώτα μια αξιολόγηση αυτών που έχουν ε, εγκριθεί, νομοθετηθεί, για να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχει αυτό αντίκτυπο στον αριθμό ε, των εικονικών εταιριών και ε, την κλίμακα της χρησιμοποίησής του Η μελέτη πάντως ε, ε, επικεντρώνεται στις ε, εικονικές εταιρείες εντός της Ένωσης. Σας ευχαριστώ, ο Ραμόν. ναι, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, διότι ξέρω ότι άργησα. Είχα, ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση, δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Θα ήθελα να ξέρω, εάν στην έρευνά σας για αυτές τις ε, εικονικές εταιρείε, τις εταιρείε φαντάσματα όπως λέμε εμείς, ε, εξετάσατε το θέμα του, του Γιβραλτάρ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρωτόκολλο στα πλαίσια του Brexit και ένα από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας με τον ΕΒ Βασίλειο και, την Ισπανία είναι αυτό. Ε, υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας για, την, για μια πιο στενή ε, συνεργασία, ελπίζουμε, ε, μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας ε, στο φορολογικό τομέα. Και μια πολύ μεγάλη διτερότητα αυτής της περιοχής. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 25.000 ανθρώπων, έτσι. Πριν από λίγο καιρό υπήρχαν 23.000 εταιρείε εκεί και αυτά βεβαίως, ε, αυτές οι εταιρείε ε, ανταποκρίνονται ακριβώς σε αυτά τα χαρακτηριστικά που πάτε εσείς. Καθόλου ε, οι πολύ λίγοι ε, εργαζόμενοι, καθόλου η πολύ λίγη δραστηριότητα και καθόλου η πολύ λίγη φυσική παρουσία. Ε, έχετε εξετάσει στη μελέτη σας την περίπτωση αυτή, αυτό τον ειδικό, πώς να το πω, χώρο, ε, αυτό, εμπασχεπτώσει, το μέρος, που ονομάζεται Γιβραλτάρ και που βρίσκεται στην Ισπανία. Όχι, όχι, για να απαντήσω σύντομα, όχι, δεν, δεν μελετήσαμε το Γιβραλτάρ. Εμείς εξετάσαμε, ε, εξετάσαμε ε, κράτη-μέλη της Ένωσης χωρίς υπερπόντια ε, εδάφη διαμερίσματα αλλά η μελέτη που παρουσιάστηκε πέρυσι και την οποία εμείς, την, παραπέμπουμε, που έκαναν επίσης συνάδελφοι του EPRS, που ε, εξέτασε ε, συγκεκριμένα αυτά τα εδάφη, θα το βρείτε κάπου σε μια υποσημείωση, εκεί που μιλάμε ε, για το γεωγραφικό πεδίο που θέλουμε να καλύψουμε και μιλάμε για τον αποκλεισμό των υπερπόντιων εδαφών. Βεβαίω για αυτού του τρει δείκτε, εάν εφαρμοστούν αυτοί οι τρει δείκτε, ε, σε Πολλά υπερπόντια εδάφη και διαμέρισματα ε, προφανώς ε, θα δούμε πολύ υψηλές ε, ε, πολύ υψηλή ισχύ αυτών των κριτηρίων για τις ξένες εταιρείε, για τις άμεσες εξωτερικές επενδύσεις, για το, τις εταιρείες ειδικού σκοπού. δηλαδή σίγουρα σχετίζονται με αυτές τις χώρες, ε, αυτές τις δραστηριότητε. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους ε, που είναι παρόντες αν έχουν περαιτέρω ερωτήσει. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Στην περίπτωση αυτή να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, της προσκεκλημένης μας που ήλθαν εδώ σήμερα και που κατέβαλαν τόσο μεγάλη προσπάθεια ε, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών και να ζητήσω συγγνώμη για το γεγονό ότι σήμερα δεδομένων ανελειμμένων υποχρεώσεων βρέθηκαν να κάθονται μπροστά σα και να έντρανα σε μια κατάσταση που δεν έχω ξαναζήσει να πω την αλήθεια. Τρία άτομα μόνο να έχουμε μαζί μας σε όλη τη συνεδρίαση. Και να ευχαριστήσω και όλους εκείνους ε, που παρακολούθησαν μέσω web streaming την ε, συνεδρίασή μας να επισημάνω ότι υπάρχει το EPRS σε μια φανταστική εφαρμογή την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε από το App Store και εκεί μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της σημερινής συνεδρίασης ε, είναι πραγματικά εξαιρετική η εφαρμογή. Πιο διαφανής δεν γίνεται να είναι οι συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξαιρετικό πιστεύω. Και μην ε, αμελήσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ε, να σας ευχηθώ καλό απόγευμα και λήξη της συνεδρίασης.